Welcome back to you all. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε πάλι στη συνεδρίασή μας. Περιμένουμε ακόμα μερικούς συναδέλφους προκειμένου να κάνουμε τη συζήτηση που προβλέπεται στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Οικονομικό Έτος 2020. Η συνάδελφος Γκαρθιαρμπάλα είναι παρούσα, επομένω μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και αντί να ξεκινήσουμε με το τμήμα 3, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα τμήματα για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προχωρήσω περιμένοντας. Πάρα πολύ σύντομα. Σχετικά με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών, λέει η κυρία σαπάλ, έτσι ώστε να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες αποκατάστασης των περικοπών τις οποίες έχει προβλέψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ελπίζω ότι στις συναντήσεις τις οποίες κάναμε μέχρι τώρα και στις μελλοντικές τις οποίες θα έχουμε και πριν το τέλος της εβδομάδας να μπορέσουμε να λύσουμε τις διαφορές που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελπίζω ότι η επικοινωνία εδώ έχει σταθεί λίγο δύσκολη μέχρι τώρα και περιπλέκεται και λόγω του Brexit φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Προϋπολογισμών στις προηγούμενες συνεδριάσεις αποφάσισε να αποκαταστήσει πλήρως ουσιαστικά την ανάγνωση την οποία είχε κάνει το ίδιο το προϋπολογισμό και να αποκαταστήσει τους αριθμούς τους οποίους είχε περικόψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν τώρα ορισμένες τροπολογίες τις οποίες ονομάζουμε τεχνικού τύπου στην ουσία θα προετοιμαστούμε για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν, δηλαδή ε, το Brexit, το τι θα γίνει μετά από, το, ε, από τις 31 Οκτωβρίου είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει κατά πολύ ε, στη συνέχεια και επίσης υπάρχει και μια διόρθωση η οποία θα πρέπει να γίνει για τα έξοδα των βουλευτών οι οποίοι δεν έχουν επανεκλεγεί ε, και το συνολικό ποσό το οποίο χρειαζόμαστε είναι υψηλότερο από αυτό το οποίο είχαμε στην διάθεσή μας. Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Τώρα για τους προϋπολογισμούς των υπολείπων κοινοτικών οργάνων. Έχουν κατατεθεί ορισμένες τροπολογίες και υπάρχει συνένεση επίσης για την αποκατάσταση, για την επιστροφή ε, στην αρχική πρόταση και ε, απομάκρυνση των περικοπών τις οποίες είχε καταλήξει, στις οποίες είχε καταλήξει το Συμβούλιο. Εμείς εδώ βασιζόμεθα στην ανάγνωση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποκατάσταση των αριθμών για την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, για την Επιτροπή των Περιφερειών και για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο εδώ. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε στην ουσία καταλήξει σε αρκετά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις έφτασε και ο κύριος Φερνάντες, μήπως να σας δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα την παρουσίαση της ε, κυρίας Γκαρθιά Θαμπάλ Ρουμπιάλ για τα υπόλοιπα τμήματα. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έλεγα πάντα ότι οι προπολογισμοί θα πρέπει να είναι αυστηροί κατά την εφαρμογή τους. Έτσι και με τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μπορούμε να επιτελούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νομοθετικό μας έργο. Συμφωνούμε με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Συμφωνούμε επίσης με την εισηγήτρια για τα υπόλοιπα τμήματα του προπολογισμού. Συμφωνούμε επίσης με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέρα από αυτό το ζήτημα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι στα πλαίσια των συμφωνιών και ιδίω του Gentleman Agreements υπάρχουν συγκεκριμένε ρήτρε τι οποίε πρέπει να τηρήσουμε. Αυτέ θέλουμε να προσπίσουμε σε σχέση με το Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμφωνία αυτή να μην αποδυναμωθεί από το Συμβούλιο. Ο στόχος μας είναι εδώ πέρα να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα το έργο μας, να έχουμε το απαραίτητο επίπεδο διαφάνειας και όπως σας είπα όλα τα όργανα θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να αποκριθούν στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Καταλαβαίνετε ότι όταν τα όργανα δεν έχουν τα απαραίτητα αυτά μέσα, τότε αυτό οδηγεί σε πολύ σημαντικές δαπάνες, τόσο διοικητικές όσο και επιχειρησιακές. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τα επίπεδα τα οποία θέλουμε για τον προπολογισμό των οργάνων αυτών. Ένα 93% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Αυτό δεν το βλέπουμε καθόλου σε εθνικό επίπεδο. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί μόνο τα απόδειξη ότι η εργασία που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί προστιθέμενη αξία. Οτιδήποτε καταγράφεται στον προπολογισμό αντιστοιχεί τελικά σε μια προστιθέμενη αξία η οποία αποφελεί τελικά τα ίδια τα κράτη-μέλη και του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε. Ο κύριο Σαστέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την εργασία των εισηγητών μας. Θεωρώ ότι η συναντική αυτή εργασία που έχει γίνει είναι υποδειγματική και οι συζητήσεις και οι επαφές που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικές προκειμένου να καταφέρουμε να αποσαφηνίσουμε συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπόθηκε και κατά την παρουσίαση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε στα πλαίσια της συζήτηση αυτής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά είχε αρχίσει να παρισφρεί στην κατάρτιση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τρεις γραμμές του προπολογισμού. Για δύο από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πρόβλημα χάρη στην εργασία που έχει κάνει ο εισηγητής μας, αλλά για την τρίτη γραμμή του προπολογισμού που εκκρεμεί ακόμα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την εργασία μας. Έχουμε σημαντικές τροπολογίες τεχνικής φύσης που αντιστοιχούν σε εξελίξεις που είχαμε το 2019 σε σχέση με το Brexit αφενός και αφετέρου σε σχέση με τις εκλογές και την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα θελήσαμε να επιστρέψουμε στον αρχικό προπολογισμό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακτώντας βασικά τις περικοπές που είχαν γίνει στο παρελθόν, ερχόμενοι σε συνεργασία περισσότερο με το Συμβούλιο. Έπειτα είχαμε κάποιες εξηγήσεις που μας δόθηκαν από τα υπόλοιπα όργανα, πολύ σαφείς εξηγήσει για το πώς θα χρησιμοποιούσαν τα ποσά τα οποία απαιτούσαν και μετά τις εξηγήσει αυτές εμείς καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να ανακτηθούν τα ποσά αυτά και να επιστρέψουμε στα αρχικά προτινόμενα ποσά. Και κατά αυτόν τον τρόπο καταλήξαμε σε μια ομοφωνία μεταξύ των διαφορετικών εισηγητών και σχεδόν εισηγητών σε σχέση με τα συμπεράσματα αυτά τα οποία σας παρουσίασε και ο εισηγητής μας. Αυτά όσον αφορά τον προπολογισμό των υπολείπων τιμιωάτων. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κύριο Αντρέσεν. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πολλές φορές διήστανται οι απόψεις σε σχέση με τους διάφορους τίτλους του προπολογισμού που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους τομείς. Για τους πράσινους πάντως το ζήτημα είναι θεσμικό και δημοκρατικό ουσιαστικά. Δεν θα πρέπει να, να περικόπτουμε τον προπολογισμό που προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για αυτό το λόγο στηρίζουμε πλήρως την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κούνσε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μια και είμαι εντελώ καινούριο εδώ στην διαδικασία και στην κατάρτιση του προπολογισμού, θα ήθελα να μην εκφράσω οποιαδήποτε άποψη. Θα ήθελα να απόσχω. Και είναι ακόμα πολύ πρώιμη φάση για να μπορώ να έχω μια άποψη από αυτόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόντσα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι με την τροπή της συζήτησης ως τώρα. Το ΕΣΥΑΡ έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα Και αυτό έχει να κάνει με την ρεαλιστική προσέγγιση που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε για το 2020. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Άλλα σχόλια για τα άλλα τμήματα, μήπω. Έχετε το λόγο. Το όνομά, το όνομά μου το προφέρετε τώρα πια. Τα καταφέρνετε, σιγά σιγά. Μία εβδομάδα σας δίνω. Και τώρα θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Εσείς το όνομά μου το δικό μου το λέτε. Θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψε την ερχόμενη εβδομάδα. Ας περάσουμε στο προκειμένο τώρα. Ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή γιατί πιστεύω ότι αυτό που προτείνεται είναι το ελάχιστο που οφείλει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να υπερασπιστεί μέχρι τέλους ότι πρέπει να πάψουν και επομένως να αρθούν οι περικοπές οι οποίες εισηγήθηκε η Κομισιόν να γίνουν. Πιστεύω ότι αυτό δεν αρκεί. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλει να είναι συνεπές με τον εαυτό του, με δεδομένο ότι από το Συμβούλιο θα έχουμε μία επίμονη ε, προσέγγιση στη λογική των περικοπών, όχι μόνο στον προϋπολογισμό για το 2020, αλλά και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προετοιμαστεί με θετικές προτάσεις για ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό, ο οποίος όχι απλώς να μην έχει περικοπές, αλλά, αλλά να έχει και αυξήσεις σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας, όπως είναι κλιματική αλλαγή ή πολιτικές συνοχής. Και πρέπει να αγγίξουμε με δική μας πρωτοβουλία και το θέμα της αύξησης των ιδίων πόρων. Είναι κρίμα προτάσεις όπως αυτές που ετοίμασε η Επιτροπή Μόντι να μένουν στο κάτω μέρος του τελευταίου συρταριού και της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Okay, this, this was... Μάλιστα. Αυτό ήταν το τρίτο τμήμα. Αλλά είμαστε ακόμα στα υπόλοιπα τμήματα. Θέλετε να πάρετε το λόγο για τα άλλα τμήματα ή για το τρίτο τμήμα. Ε, πραγματικά ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ απόλυτα με τον αγαπητό φίλο συνάδελφο τον Τζοζέρ Μαλέρ Φερνάντε είναι ένα κοινωνικό επενδυτικό προπολογισμό που το 93% των δαπανών του κατευθύνεται προ την ανάπτυξη. Και αδικείται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν κάποιοι συστηματολογούν και λένε ότι οι προπολογισμοί τη είναι νεοφιλελεύθεροι, ότι είναι προπολογισμοί λιτότητα, ότι είναι προπολογισμοί περικοπών. Ταυτόχρονα συμφωνώ ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αυξηθεί από μόνο του. Πρέπει να συνεισφέρουμε. Εμεί ακριβώ επειδή θέλουμε ένα πιο ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό προπολογισμό, στηρίζουμε την άποψη ότι ο προπολογισμό πρέπει να ενισχυθεί αυξάνοντα τη συνεισφορά των χωρών μελών στο 1,3. Και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε και την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσουμε και τον κοινωνικό και τον αναπτυξιακό προπολογισμό. Και ένα ιδιαίτερα σημαντικό για μα Πολλέ φορέ σε αυτήν την αίθουσα σχετικά με τη συζήτηση με τον προπολογισμό είπαμε ότι ένα προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται σε αρχέ και αξίε πρέπει να συνδέεται και με το κράτο δικαίου. Δηλαδή, χώρε όπου και αν βρίσκονται αυτέ που δεν εφαρμόζουν το κράτο δικαίου, που δεν εφαρμόζουν ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από του Ευρωπαίου πολίτε. Και κανένα Ευρωπαίο πολίτη δεν είναι διατεθειμένο να χρηματοδοτεί αυτέ τι χώρε. Έχουμε όμω το χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Τουρκία, που παραβιάζει το κράτο δικαίου εντό τη χώρα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα επιτίθεται σε όλε τι χώρε, τι γειτονικέ χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και Τουρκία. Και συνεχίζουμε. Okay, I will finish only one second. I... Και συνεχίζουμε let, να me, let me insist, we, were on other sections. Επιμένω, λέει ο Πρόεδρος, ότι είμαστε σε άλλα τμήματα, συζητάτε άλλο θέμα, άλλο τμήμα. Να ακολουθούμε, αν θέλετε, τη σε σειρά. Ναι, μια γενική άποψη εξέφρασα, ναι, ναι, ναι, αλλά για το τμήμα 3. Η κυρία Χόλμαϊρ. Μόνικα, Μόνικα. Sorry, I was asking Ναι, συγγνώμη. Μία ερώτηση έκανα. Ναι, όχι, ζητώ, ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Πρόεδρε. Δεν ήμουν προσεκτική. Συνάδελφοι. Καταρχάς, για τον προπολογισμό της Επιτροπής και τα κοινωνικά ζητήματα που τίθενται σε αυτόν. Σας έστειλα μια συμβιβαστική πρόταση και υπήρχε παρεξήγηση για το κατά πόσον ήταν συμβιβασμό του ΕΛΚ. Όχι, είναι συμβιβασμό γενικά, όχι του ΕΛΚ. Είναι λοιπόν έργο τη εισηγήτρια για να υπάρξει συμβιβασμό μεταξύ των προτάσεων όλων των πολιτικών ομάδων. Όχι να υποβληθεί κάτι από πλευρά μόνο του ΕΛΚ. Κατά δεύτερον. Στα πλαίσια της πρότασης αυτής, στο 1α, όχι μόνο χρειαζόμαστε τα περιθώρια που προβλέπονται, αλλά θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και άλλα ειδικά εργαλεία, ειδικά μέσα. Και μάλιστα μεγάλη χρηματική κλίμακας, το οποίο στην τελική ανάλυση θα οδηγήσει όχι μόνο μην έχουμε περιφέρεια, αλλά και το εργαλείο ευελιξία και το τις παγκόσμιες δεσμεύσεις θα πρέπει να τα δεσμεύσουμε για το 3 τις αποδεσμεύση Στο 1β τώρα, παρόμοια κατάσταση, γιατί χρειαζόμαστε τα επιπλέον εργαλεία για το πρόγραμμα Yay, το Youth Employment Initiative. Θα πρέπει να προταθούν λοιπόν επιπλέον εκατομμύρια γιατί η βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφώς χαμηλότερη από ό,τι την περσινή. 233 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, 116 φέτος. Και αυτό δεν θα εμφανιστεί στο πουδουπού, αλλά θα ενταχθεί στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κτλ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα παρουσιάσετε το θέμα της ε, νεανικής ενεργείας εδώ. Αυτό το πρόγραμμα έχει βάση χρονική διάρκεια 2-3 ετών. Σε τελική ανάλυση λοιπόν, αυτά που γίνονται σε βάση ετήσια δεν μπορούν να επεκταθούν σε μεγαλύτερο σε χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω 33 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτά τα 53 εκατομμύρια δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν πέρσι. Και αν θέλουμε να συνεχιστούν τα προγράμματα αυτά, θα πρέπει στο πλαίσιο του επόμενου που να δούμε πώς θα μπουν στο ESF, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Έχουμε κάποιο περιθώριο που περισσεύει γιατί οι νομικά προδιαγραμμένες ε, τα χαρτοφυλάκια για τα κράτη μέλη έχουν ήδη προδιαγραφεί, άρα δεν έχουμε περιθώριο. Έχουμε όμως στο live ε, ένα περιθώριο και ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού μπορεί να απορροφηθεί αυτό το περιθώριο για να μπορέσουμε να καταθέσουμε επιπλέον προτάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων. Στο τρίτο τμήμα έγιναν πολλές προτάσεις, κυρίως από σοσιαλιστές και δημοκράτες, μεγάλη, μεγάλης κλίμακας. 122 εκατομμύρια επιπλέον στο ε, τμήμα 4. Δεν θα μας ε, παραμείνει τίποτα, δεν θα έχουμε περιθώριο για τίποτα άλλο, γιατί από την αναπτυξιακή βοήθεια δεν μένει τίποτα ποτέ. Πάντα θέλουμε να ενισχύσουμε την αναπτυξική βοήθεια και ακριβώς αυτό το ερώτημα ε, έθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού μπορούμε να απορροφήσουμε περαιτέρω κονδύλια και πού δεν υπάρχει ποσόστοση απορρόφησης. Ακούστηκαν διάφορες επιθυμίες από, τα, από τις πολιτικές ομάδες. Στο πέμπτο τμήμα, τα είπαν οι συνάδελφοι, δεν έχω να διευκρινίσω τίποτα. Έχουμε ένα περιθώριο. Κοιτώντα λοιπόν την συνολική συζήτηση για το τελευταίο έτο, θα ήθελα να τονίσω το εξή. Δεν υπάρχουν χρήματα τα οποία να υπάρχουν σε κάποιο ε, χρηματοκιβώτιο. Δεν υπάρχουν χρήματα. Όλα αυτά που αποφασίζουμε είναι δεσμεύσει πληρωμών που κάποια στιγμή θα πρέπει να κατατεθούν στο μέλλον. Στην παρούσα λοιπόν φάση, στο δεύτερο που, που δεν θα έχουμε μόνο το 2020, αλλά και τα N+, 2021, 2022 και 2023. Αυτό σημαίνει ότι αν θέσουμε παράλογα προγράμματα, δεν θα έχουμε στο νέο που που χώρο για νέα έργα, γιατί όλα αυτά θα μπουν στο πρώτο έτος. Ο κ. Λεβαντόφσκι το γνωρίζει το πρόβλημα και από το παρελθόν. Παλιά είχαμε το νήσιν 2, τώρα θα έχουμε και νήσιν 3. Αυτό λοιπόν θα επιδεινώσει τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε κάποια χρήματα για την τελευταίο έτος. Για παράδειγμα το μέσο ευελιξίας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα περιθώρια. Θα πρέπει να βάζουμε το καθολικό περιθώριο για τις δεσμεύσεις για όλα αυτά τα θέματα για το κλίμα, για θέματα ψηφιοποίησης. Θα πρέπει επίσης να πείσουμε και το Συμβούλιο και να σας πω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε το Συμβούλιο για το 15-3. Όποιος ήταν την προηγούμενη φορά εκεί και είδε τι αντίσταση είχαμε για το 15-3 από το Συμβούλιο, θα ξέρει ότι ε, λε και δεν τα ξέραν όλα αυτά όταν τα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Φυσικά και τα ήξεραν. Προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε κάποιο περιθώριο και στο 15.3. Η άποψή μου είναι η εξή, ότι το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε για δημοσιονομική πειθαρχία σε ό,τι αφορά το θέμα της έρευνας και προκειμένου να μην συνεχίζονται προγράμματα τα οποία δεν τα πηγαίνουν καλά, αλλά να συγκεντρώνονται τα κονδύλια και να δαπανώνται για νέα καλά έργα. Αυτό είναι η ιδέα πίσω από το 15.3. Αν το απορρίψει το Συμβούλιο το 15.3, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα θεωρήσουν ότι τι δεν τα κάνουμε όλα αυτά τα χρήματα και γιατί τα μαζεύουμε αφού δεν έχει καλό στόχο. Ελπίζω λοιπόν αυτό το επιχείρημα να πείσει το Συμβούλιο. Αλλά έχω μία έκκληση να απευθύνω προς τους συναδέλφους, το είπα και σήμερα το πρωί προς τους συντονιστές. Η πρόταση την οποία κάνω σίγουρα είναι μια συμβαστική πρόταση. Το ΕΛΚ, να σας το πω ξεκάθαρα, θα ήταν πολύ χαμηλότερα από την πρόταση αυτή. Το λέω ξεκάθαρα γιατί όπως είπε ο συνάδελφος Γκάιρε από τους σοσιαλιστές, ε, οι τελευταίες ε, εμπειρίες μα στη συνδιαλλαγή ήταν πολύ αποτελεσματικέ, πολύ απογοτευσικές. Και οι τίτλοι στι εφημερίδες για τα αποτελέσματα που θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να τα προωθήσουμε στην κοινή γνώμη παρουσιάστηκαν με άσχημο τρόπο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρουσιάστηκε ότι και καλά οι ευρωβουλευτέ θέλουν να τα ξοδέψουν όλα, να τα σπαταλήσουν όλα. Θα ήθελα να σα προειδοποιήσω λοιπόν να μην γίνει τέτοια συζήτηση. Το τελευταίο εργαλείο, contingency margin, 900 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν θα έλεγα να μην το αγγίξουμε και αυτό για λόγους ουσίας, γιατί την επόμενη περίοδο θα δούμε ε, πώ θα φτάσουν, για παράδειγμα, όλο και πιο μεγάλη αριθμή μεταναστών στα σύνορά μα. Είμαι απολύτω σίγουρη ότι θα έρθει μια συζήτηση για το πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε πρόσφυγε, πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε άτομα τα οποία διαφεύγουν με διάφορα εργαλεία, με διάφορα μέσα. Αυτό λοιπόν αυτόματα θα μπει στον προπολογισμό μα. Αυτό σημαίνει ότι από κάπου θα πρέπει να έχουμε και ένα περιθώριο στον προπολογισμό αυτό, προκειμένου τα ε, εργαλεία τα οποία έχουν προβλεφθεί καλά. Αυτό το contingency margin, αυτό το περιθώριο της ανάγκης λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει. Αυτά τα 900 εκατομμύρια δεν τα ακούμπησα στην συμβιβαστική πρόταση από πλευράς ΕΛΚ και από πλευράς ε, των, της οπτικής των συναδέλφων μου, έχω ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που θέλαν. Προσπάθησα να καταθέσω μια συμβαστική πρόταση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό και είναι διχασμένο το κοινοβούλιο, αυτό σε τελική ανάλυση θα σημαίνει ότι έχουμε de facto χάσει ήδη. Αν κατέβουμε με διαφορετικές προτάσεις ή για παράδειγμα αν δεν είναι σε ισχυρή θέση η συγγήτρια να ξεκινήσει την Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να αντιληφθείτε το εξή. Η πρόταση που κάνουμε για το 1α, να σας πω ότι οι προτάσει αυτέ είναι 10 πλάσιες σε σχέση με το 2018 και 20 πλάσιες σε σχέση με το 2017, σε σχέση με την πρότασή μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω. Αν θέλει κάποιο να μου εξηγήσει ότι θα πρέπει να πάμε πιο υψηλά επίπεδα, να ξεπεράσουμε περι... ακόμα πιο πολύ τα όρια αυτά, θεωρώ ότι θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να ενταχθούμε στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν ε, αντιδρώ βάση των επιθυμιών μου. Αν ήταν οι επιθυμίε μου η βάση, θα είχα πολλέ επιθυμίε να εκφράσω. Κινούμε στο πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθώ, στο πλαίσιο του πουδουπού, σε ό,τι αφορά τις διάφορες ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και είναι πολύ διαφορετικές, ε, να σας πω, από ομάδα σε ομάδα Γι' αυτό λοιπόν ε, σας παρακαλώ ως εισηγητρία δώστε μου την ευκαιρία να πετύχουμε ένα καλό συμβασμό και να έχουμε μια κοινή πρόταση ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιτρούο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή Μόνικα, ευχαριστώ για το κείμενο που προτείνεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμά ε, επιθυμούμε να υπάρξει μια κοινή θέση του Κοινοβουλίου η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο θα είναι δύσκολη. Ευχαριστώ επίσης και για τον διάλογο τον οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες. Σίγουρα η πρόταση είναι καλύτερη από την αρχική, έχει υπάρξει πρόοδος για την απασχόληση των νέων και για το κλίμα. Εμείς ως σοσιαλδημοκράτες θεωρούμε ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν έχουμε καταλήξει τον καλύτερο συμβιβαστικό τρόπο να συνεχίσουμε είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να είμαστε σοβαροί και να χρησιμοποιήσουμε κάποια αποθηματικά περισσότερο. Υπάρχουν 904 εκατομμύρια ευρώ σε αποθεματικό για έκτακτες καταστάσεις. Εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το 100% το είπα και σήμερα το πρωί. Το συζητήσαμε και στο μεσημεριανό διάλειμμα. Πρέπει να κρατήσουμε κάποια από τα αποθέματα αυτά αλλά από το να χρησιμοποιήσουμε 904 ή να μην χρησιμοποιήσουμε κανένα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η κατηγορία 5 είναι οι διοικητικές δαπάνες. Ξέρουμε ακριβώς ποιες θα είναι το 2020. Γιατί να κρατήσουμε λοιπόν 672 εκατομμύρια εδώ στο αποθεματικό. Μπορούμε για την κατηγορία 2 να έχουμε κάποιο αποθεματικό και μάλιστα ε, προτείναμε αύξηση του ποσού αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το αποθεματικό για την κατηγορία 5. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ένα τμήμα τους. Είπες ότι θες έναν προϋπολογισμό βιώσιμο. Η σοσιαλδημοκρατία όμως θέλει και ένα πλανήτη βιώσιμο. Ε, η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα πρέπει να τους θέσουμε μπροστά των αντιθέσεών τους. Όλα τα είπαν χτες στη Νέα Υόρκη, όλοι είπαν ότι είναι η προτεραιότητα είπαν ότι καίγεται ο πλανήτης. Έχω εδώ το κείμενο του ΟΣΑ που λέει ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από την ύφεση. Ήμουνα με τον Μπρινό Λεμέρ την Πέμπτη, συνάντησε τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας και είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δημοσιονομικά μέσα και όχι μόνο τα νομισματικά. Ε, και συζήτησαν Γερμανοί και Γάλλοι και είπαν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δημοσιαναμικά μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε. Και εμείς δεν θα το κάνουμε, θα το κάνουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια από αύριο το πρωί έτσι ώστε με αξιόπιστο τρόπο να καταλήξουμε σε ένα προϋπολογισμό αξιοπρεπή και βιώσιμο αλλά και να προστατεύσουμε τον πλανήτη, να δημιουργήσουμε θέσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε να συνεχίσουμε στην διαπραγμάτευση να είμαστε μέρος. Η κυρία Αμά. Ευχαριστώ. Από πλευρά των Ρινιού. Εγώ είμαι νέα βουλευτής, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τον διάλογο ο οποίος προηγήθηκε ανάμεσα στις ομάδες. Ευχαριστώ ε, την εισηγήτρια, την ευχαριστώ για τη συνεργασία που μας ακούει. Δεν έχουμε καταλήξει βέβαια ακόμα, θα συνεχίσουμε για μία ή δύο εβδομάδες ακόμα. Πάντως οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για τις μικρομεσαίες, για το Εράσμος, για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, για το Europol, όλα αυτά είναι θετικά. Είμαστε πολλοί νέοι βουλευτές που προσπαθούμε να ακούμε τους ε, βουλευτούς πολίτες μας οι οποίοι μας λέγουν ότι θα πρέπει να προσέξουμε επειδή είμαστε για πρώτη φορά εδώ. Ε, οι δύο βασικές προτεραιότητες στις οποίες εμένουμε είναι η νέα οικονομία, η οποία ανασέβεται φυσικά το περιβάλλον και δεύτερον να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ρήξης ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Για το πρώτο θέμα θα πρέπει να αποδείξουμε ότι ακούμε τους συμπολίτε μας, δεν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιήσουμε όλα τα περιθώρια τα οποία έχουμε για το κλίμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε να επιστρέψουμε 8 δις Τώρα είμαστε πραγματικά στο, τελευταίο, στο τελευταίο έτος αυτού του οικονομικού κύκλου. Γνωρίζουμε ακριβώς τι έχουμε μπροστά μας. Το πρόβλημα είναι περισσότερο η έλλειψη απορροφητικότητας, η μη απορρόφηση συγκεκριμένων πιστώσεων. Τώρα για το, για το ρήγμα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Και εδώ τίθεται θέμα απορροφητικότητα στην Ανατολή. Θα πρέπει η τεχνική συνδρομή ε, να βοηθήσει στην απορρόφηση των διαθέσιμων πιστώσεων στην Ανατολή. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσει ο διάλογος, πρέπει να καταλήξουμε σε μια θέση η οποία ελπίζω να είναι η πιο κοντινή στις επιθυμίες των πολιτών μας. Ο κύριος Αντρέσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στον Μάνφρετ Βέμπερ, ο οποίος σήμερα σχολίασε τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, όπου είπε ότι ε, είναι πραγματική η επίγουσα αυτή η ανάγκη που έχει προκύψει όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται λοιπόν ε, η ε, δέουσα ηγετική στάση από τους υπεύθυνου. Εμείς συμφωνούμε με αυτό ως πράσινοι και θεωρούμε ότι όντως θα πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με τον προπολογισμό του 2020. Τι σημαίνει αυτό, να κινητοποιήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε στον προπολογισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που θα καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή. Και βέβαια δεν μπορούμε να επιλύσουμε μόνο μέσω του προπολογισμού του 2020 την κλιματική αλλαγή, μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι μια αρχή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια αποθεματικά τα οποία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτό δεν το λέει μόνο ο Μάντφρεντ Βέμπερ, το λένε και πάρα πολλοί άλλοι ότι πραγματικά αντιμετωπίζουμε μια έκτακτη κατάσταση αυτή τη στιγμή, μια ιδιαίτερα επίγουσα κατάσταση. Οι επιστήμονες μας λένε ότι τώρα πρέπει να λάβουμε δράση. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια ηγετική θέση όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μέσω της χρηματοδότησης. Μέσω της χρηματοδότησης περισσότερων προγραμμάτων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ ισχυρή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη πραγματεύση που θα έχει με το Συμβούλιο. Νομίζω πάντως ότι ε, θα πρέπει να θέσουμε, αν θέλετε, μεγάλα σχέδια μπροστά μας και να μην περιοριστούμε απλώς ε, σε κάποια βραχυπρόθεσμα προγράμματα όπως είχαμε κάνει στο παρελθόν. Λοιπόν, πρέπει να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα προς το Συμβούλιο ότι ήδη από τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούμε με έναν ιδιαίτερα απόλυτο και αποφασιστικό τρόπο και με τη βοήθειά σας ε, κυρία Συγήτρια βλέπουμε ότι η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας αυτή τη στιγμή είναι μια πρόταση που θα μπορέσει ενδεχομένως να κερδίσει και άλλες πολιτικές ομάδες, να μην έχει δηλαδή μόνο την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Βέβαια θα πρέπει να πραγματιστούμε λίγο περισσότερο την πρόταση αυτή, προκειμένου να έχουμε με το μέρος μας όσο δυνατόν περισσότερες πολιτικές ομάδες. Πρόεδρος, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Λεβαντόφσκι. Σας ευχαριστώ. Συζητάμε σήμερα την αιτήσια δημοσιονομική διαδικασία όπου βλέπουμε βέβαια να παίζεται το σύνηθες παιχνίδι, περικοπές από το Συμβούλιο, απόπειρες αποκατάστασης κάποιων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το καθεξής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ε, κάποιες γραμμές του ετήσιου προπολογισμού που είναι σημαντικότατες και για το γενικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Μόνικα Χολμάιρ αναφέρθηκε και στις γραμμές αυτές. Οι γραμμές αυτές του προπολογισμού έχουν να κάνουν με την ευελιξία και έχουμε το περίφημο άρθρο 15 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Μέχρι το 2018 είχαμε κάποιες αποδεσμεύσεις κονδυλίων. Οι αποδεσμεύσεις ήταν απλώς αποδεσμεύσεις και τίποτα παραπάνω. Τώρα με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε το σημείο 2 που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά τα οποία έχουν αποδεσμευτεί υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχουμε και ακόμα ένα πιο σημαντικό άρθρο, το άρθρο 15 παράγραφος 3, που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά που έχουν αποδεσμευτεί στον τομέα της έρευνας. Νομίζω λοιπόν ότι σε επερχόμενε διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να τονίσουμε την πτυχή αυτή με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μουρισάν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις κι εγώ. Πρώτον, θα πρέπει τώρα να αποφασίσουμε για το ποια θα είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό, αλλά αυτή τη στιγμή σε αποφασίσουμε κάτι θα πρέπει να περιέλθουμε σε πολύ σκληρέ διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, άρα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και θα είμαστε ισχυροί στι διαπραγματεύσει αυτές αν είμαστε όντω ενωμένοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να νικήσουμε στο προπολογισμό του 2020, γιατί όταν θα περάσουμε έπειτα στη διαπραγμάτευση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η φάση θα είναι ακόμα πιο αποφασιστική και αν διχαστούμε στον προπολογισμό του 2020, στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε δηλαδή με το Συμβούλιο, θα αποδυναμώσουμε πάρα πολύ την διαπραγματευτική μας θέση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας. Ο εχθρός δεν βρίσκεται στην αίθουσα αυτή, ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ πέρα όλοι μας ουσιαστικά θέλουμε ένα προπολογισμό που να χρηματοδοτεί με το σωστό τρόπο τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην νεολαία, την έρευνα, την ανάπτυξη, άλλοι στην κλιματική αλλαγή. Πάντως όλοι μας συλλογικά θέλουμε να υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση και η καλή δαπάνηση των χρημάτων αυτών. Από την άλλη όμω, στο Συμβούλιο έχουμε απλούς λογιστές οι οποίοι προχωρούν σε πολύ σημαντικές περικοπές χωρίς να διέπονται αυτές από κάποια πραγματική πολιτική ανάλυση της κατάστασης. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, να είμαστε ρεαλιστές. Πολύ συχνά, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων που έχουμε το Συμβούλιο, καταφέρνουμε να περάσουμε τη δική μας τη θέση αν έχουμε πάρει με τη δική μας την πλευρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσα εισηγητήσε τον προπολογισμό του 2018, είδα ότι με αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η θέση μας θα είναι πολύ πιο επιτυχή, σαν ρεαλιστική και μετριοπαθής. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια ευαισθησία αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο ιδιαίτερα έντονη ενώπιον των επερχόμενων διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Βλέπουμε ότι ε, το Συμβούλιο δεν ακολουθεί πάντα τους δικούς μας στόχους. Επομένως, τα αιτήματά μας, οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι απόλυτα βάσιμοι. Θα πρέπει να πλαισιώνονται από μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Τρίτον, όσον αφορά τα περιθώρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε ένα χαμηλότερο επίπεδο για τα περιθώρια, γιατί βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος του τρέχοντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστούμε ένα αξιοσέβαστο ποσό και στα περιθώρια προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε και έκτακτε καταστάσει. Το είδαμε αυτό στο παρελθόν με τα χρήματα που χρειάστηκε να δώσουμε στην Τουρκία για την υποδοχή των προσφύγων ή στα χρήματα που χρειάστηκε να δώσουμε πολύ γρήγορα στο ταμείο το οποίο ε, συστάθηκε για την Αφρική. Νομίζω λοιπόν ότι θέλουμε προφανώ να έχουμε αύξηση του προπολογισμού. Συμφωνούμε από αυτού. Παράλληλα όμω, α κρατήσουμε το απαραίτητο επίπεδο περιθωρίων, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα του χρόνου. Άκουσα τόσο είπε ο Γάλλο συνάδελφο Λαγοκιουρού για την κλιματική αλλαγή. Προφανώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να προασπίσουμε το περιβάλλον. Αλλά μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο έτο ενό πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου που εγκρίθηκε το 2013 βάσει προτάσεων που έκανε ο Γιάννου Λεβαντόφσκι, που ήταν τότε επίτροπο. Επομένω, Όλες οι προσδοκίες που έχουμε αυτή τη στιγμή για την κλιματική αλλαγή είναι τεράστιες, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για το 2020 είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 2021-2027 δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσουμε τα απαραίτητα μέσα και τα εργαλεία τα οποία θα εξυπηρετήσουν τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή. Εν κατακλείδη να σας πω ότι θα πρέπει να απορρίψουμε άμεσα τις προτινόμενες από το Συμβούλιο περικοπές, να μην χάσουμε από αυτού πάρα πολύ χρόνο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και ευθύ αμέσω να περάσουμε στι ουσιαστικέ διαπραγματεύσει προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προγράμματα που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε συλλογικά να καταφέρουμε να προωθήσουμε έτσι τις κοινέ μας προτεραιότητες. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον, ε, την εισηγήτρια και τους εισηγητές γενικότερα και τους κοιόδης για την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει μέχρι τώρα. Για τον προϋπολογισμό του 2020 σημαντικό είναι να, να δούμε ακριβώς τι έχει προηγηθεί. Να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Δυστυχώς το Συμβούλιο, ενώ εμείς το κάναμε αυτό, το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην κατανοεί το τι συμβαίνει. Και ίσως να είναι και λάθος μας. Ίσως εμείς να κάνουμε λάθος. Όλα τα θεσμικά όργανα έχουν συμφωνήσει για τη στρατηγική 2020. Υπήρχαν στόχοι που δεν ήταν δεσμευτικοί, αλλά για το κλίμα, για την έρευνα, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Δυστυχώς δεν πετύχαμε τους στόχους μας. Και αυτό δεν είναι λάθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν δείξαμε την απαραίτητη ευελιξία. Έχουμε μια κάποια ευελιξία η οποία είναι προαπαιτούμενη για ένα τέτοιο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν δεν την επιδεικνύαμε την ευελιξία αυτή θα είχαμε καταστροφές ενώ αντιμετωπίσαμε πολλές κρίσεις όπως την της μετανάστευσης. Το Κοινοβούλιο έχει δίκιο. Το Κοινοβούλιο συνειδητοποιεί ότι δεν μπορούμε το 2020 να κάνουμε αυτό το οποίο δεν κάναμε τα τελευταία έξι χρόνια. Και θα συμφωνήσω εδώ με την εισηγήτρια λέγοντας ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έναν βασικό στόχο πρέπει να έχουν, τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό. Συνειδητοποιούμε πλήρως ότι αυτός ο προϋπολογισμός, αυτός ο μικρός προϋπολογισμός ωφελεί όλο τον κόσμο. Ακόμα και τα κράτη-μέλη τα οποία συνεισφέρουν, είναι καθαροί εισφορείς. Όλοι θα έλεγα ωφελούνται από τον προϋπολογισμό αυτό, ο οποίος παρουσιάζει μια τεράστια προστιθέμενη αξία. Ο ίδιος όμως αυτός προϋπολογισμός η δική μας πρόταση για αυτόν θα πρέπει να είναι αξιόπιστη πρόταση. Για να αντικαταστήσουμε αξιόπαστη ε, δεν θα πρέπει να ζητάμε χρήματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να απορροφηθούν. Και οι γραμμές οι προϋπολογισμού που δεν υπάρχουν, ε, δεν παρουσιάζουν δυνατότητες απορρόφησης δεν χρειάζεται να τις προτείνουμε. Και μάλιστα και πέραν του υπάρχοντος ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Συνεπώς λοιπόν θα συνεχίσουμε, θα καταλήξουμε ε, με προτάσεις NEA, ε, ενωμένοι, αλλιώς θα κάνουμε δώρο στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή προκαλεί το Κοινοβούλιο. Είδαμε ότι το 15-3 συμφωνούσαν για την ευελιξία, για τη χρήση χρήματος έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι ίδιες οι δηλώσεις του Συμβουλίου για τους νέους, για την απασχόληση των νέων. Δεν χρησιμοποίησαν λοιπόν αυτή την ε, δυνατή ευελιξία και τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν, στα θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη συμφωνούμε και συμφωνώ ε, και τους εκπροσώπους των Πρασίνων που συμπεριέλαβαν και τον πρόεδρο της πολιτικής μου ομάδας και τους στόχους που έχει για το κλίμα, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι όλοι οι ηγέτες και το ίδιο ισχύει και για τις άλλες πολιτικές ομάδες αναγνωρίζουν ότι έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή ανησυχία. Ελπίζω η ανησυχία αυτή να ληφθεί υπόψη και να γίνει σεβαστή από όλα τα κράτη-μέλη. Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι πολιτικές οικογένειες κάθε κράτους μέλους. Κάθε ένας από εμά πρέπει να πείσει, να προσπαθήσει να πείσει τους πρωθυπουργού του ότι θα πρέπει να υπάρξουν επαρκείς πιστώσεις για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γουαλμίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση. Είμαι λίγο απογοητευμένη ως νέο μέλος αυτού του κοινοβουλίου. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα για το ότι θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, αξιόπιστοι ε, και άκουσα επίσης και την άποψη που λέει ότι ο προπολογισμό είναι ένας μικρός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν παρουσιάζει πάρα πολλές δυνατότητες. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Αν αρχίζουμε τη συζήτηση με αυτή την υπεύθυνη αλλά και περιοριστική αντίληψη, δεν νομίζω ότι ποτέ θα πετύχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν είναι μια γραφειοκρατική άσκηση, δεν είναι μια τεχνική ρύθμιση είναι ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμεθα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των πολιτών μας. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και τη μηχανή ε, και τους μοχλούς για να πετύχουμε τους στόχους. Και βλέπουμε να έρχεται μια οικονομική κρίση και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Θα πρέπει να κάνουμε ε, προτάσεις επίπεδου Άκουσα επίσης για τις κοινωνικές πολιτικές, για τα κοινωνικά μέσα, για την απασχόληση των, μελ, των νέων, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι απέναντι στο Συμβούλιο και δεν θα πρέπει εμείς να αρνηθούμε, να χρησιμοποιήσουμε τον σημαντικό ρόλο που μας δίδει η δημοσιονομική πολιτική. Ο υπολογισμό του 2020 θα πρέπει να είναι μια νέα δυνατότητα έτσι ώστε να αρχίσουμε να περνάμε από μια γραφειοκρατική και δίσκαμπτη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κοινωνική και πράσινη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθω στην κλιματολογική, στον κλιματολογικό στόχο. Πραγματικά μπορεί να μας θεωρήσετε ανεύθυνος, αλλά πρώτον διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάτι το κατεπήγον για το κλίμα και δεύτερον, για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 20 θα έχουμε μία προτεραιότητα ξεκάθαρη, μία προτεραιότητα την οποία συμμερίζεται το σύνολο του Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, έχουμε τη συνέστηση των ευθυνών μας. Έχουμε μία προτεραιότητα πέραν όλων των άλλων, κλιματολογικά. Φυσικά τώρα τα τρία δις και τα λοιπά ελπίζουμε να τα έχουμε στη διάθεσή μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αποκτήσουμε. Η λογική την οποία μας παρουσιάσατε μέχρι τώρα ότι καλό θα είναι να προσπαθήσουμε γιατί το Συμβούλιο αν καταλήξουμε με πολύ φιλόδοξες προτάσεις δεν θα μας ακούσει. Αυτή η λογική εμένα δεν με ικανοποιεί και είμαι και εγώ νέα βουλευτής. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τις εκλογές της 6 Μαΐου και νομίζω ότι πρέπει να επιδείξουμε την απαιτούμενη υπευθυνότητα πηγαίνοντας στο Συμβούλιο με μία φιλοδοξία, με μία προτεραιότητα για την οποία πρέπει να δώσουμε μάχη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε όλα τα περιθώρια τα οικονομικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε ή να πλησιάσουμε στην επίτευξη του στόχου καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει τα όσα ακούσαμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφανώ ε, και καλωσορίζουμε την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ε, βουλευτών σε ό,τι αφορά τι προτινόμενε ε, τροπολογίε για τον προπολογισμό του 2020, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τα άλλα τμήματα του προπολογισμού. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γκαρδία Σιαμπάλο, ότι οι συζητήσεις ε, που έχουν γίνει είναι ήδη αρκετές και πολύ άριθμες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να επιβεβαιώσω επίσης την καλή πρόθεση και του Επιτρόπου Ότινγκερ και τη γενική μα διεύθυνση τη κυρίας Κόπμαν για να συνεχιστούν οι συζητήσει. προκειμένου να πετύχουμε συμφωνία επ' αυτών για το τρίτο τμήμα του προϋπολογισμού. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που επιβεβαίωσαν ότι στόχος του Κοινοβουλίου είναι να επαναφέρουμε τις περικοπές που έκανε το Συμβούλιο στον προπολογισμό της Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο, δεν θα κάνω σχόλια επί του περιεχομένου στην παρούσα φάση. γιατί κάθε χρόνο μόλις γίνεται η ψηφοφορία και μόλις το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ανάγνωσή του, τότε είναι η στιγμή για να κάνει σχολή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή εφαρμοσιμότητα, όπου φυσικά θα λάβουμε υπόψη και την θέση του Συμβουλίου. Αυτό θα υποβληθεί στην αρχή χάραξη του προπολογισμού αρχέ Οκτωβρίου. Πέραν τούτου, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συζήτηση για τις προτεραιότητε του 2020, καταρχάς στις 16 Οκτωβρίου στον τριμερή διάλογο και θα σας διαβεβαιώσω ότι έχει κάθε καλή θέληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει καλή συνεργασία για την ε, διαδικασία χάραξη του προπολογισμού προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία στη συνδιαλλαγή ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο που έχει η συγγήτρια για να πετύχει σε Άρα, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τη ευχηθώ καλή τύχη για την ψηφοφορία την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μήπως θέλουν να πάρουν τον λόγο οι δύο ηγητές, για να κάνουν κάποια σύντομα σχόλια. Η κυρία Χόρμαερ, δεν θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Κάντε ό,τι μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, λέει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Καταρχάς, Καταρχά για να καταλάβετε και την ψηφοφορία για την επόμενη εβδομάδα, εδώ δεν μιλάμε μόνο το θέμα, για τα θέματα ευθύνων για τις ευθύνε. Προσπάθησα να το επεξηγήσω αυτό και μάλιστα με ακριβή τρόπο σοσιαλδημοκράτες, Renew, Γκουε και οι πράσινοι υπέβαλαν τροπολογίες που είναι εκτός της νομικής βάσης. Αυτό σημαίνει ότι η νομική βάση, αν την αφήσουμε εκτός στην ψηφοφορία μας, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα κάναμε καν Θα είχε τελειώσει η όλη υπόθεση πριν πούμε μία πρόταση. Όλες οι υπόλοιπε ε, πολιτικές ομάδες, ε, αυτές μάλλον οι πολιτικές ομάδες ξεπέρασαν τα νομικά προδιαγραμμένα όρια και αυτό δεν έχει νόημα, δεν μπορώ να το υπερασπιστώ. Κατά δεύτερον, εν μέρη οι πολιτικές ομάδες έχουν διαφορετικές ε, αντιλήψεις για το πώ θα διαμορφωθούν όλα αυτά. Για παράδειγμα, συμφωνούμε για το κλίμα, αλλά δεν συμφωνούμε για τα επιμέρου. Αν τα βάλουμε λοιπόν όλα αυτά θα έπρεπε να παρατείνουμε τον προπολογισμό μα κατά 7 έτη για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα όλων των πολιτικών ομάδων. Πολύ απλά δεν γίνεται αυτό. Πολύ απλά δεν έχει βάση. Δεν στέκει. Γι' αυτό λοιπόν στου πράσινους λέω ότι είσαστε δύο δις εκτός του προπολογισμού, αν και το γεγονό παραμένει ότι μένετε μέσα στο πουδουπού. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στην κοινή λογική για τον συνάδελφο Γκουεμίν. Να πω το εξή, να διαβάσω και να καταλάβει τι ζητάμε, γιατί ε, συνήθω δεν διαβάζει κανεί αυτά. Ζητάμε λοιπόν και για τα SNEs, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλλον 20 στην καινοτομία, για την υποστήριξη 15 ε, εκατομμύρια, επιπλέον 10 εκατομμύρια και άλλα 10 εκατομμύρια για να πετύχουμε μία ανθεκτική εικόνα και βιώσιμη παροχή πρώτων υλών. 70 εκατομμύρια ζητάμε για θέματα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και το καθεξής. Ζητάμε 83 εκατομμύρια. Βελτίωση της ζωής 65 ε, εκατομμύρια. Πραγματικά παρεμβαίνουμε το θέμα είναι επίση άμα έχουμε και την απορροφητικότητα για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου απαντάει και μου λέει πως όχι, όλα αυτά δεν είναι ρεαλιστικά. Πιέρ, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λες, αλλά το πέμπτο τμήμα περιλαμβάνεται στο contingency margin, αυτό στο περιθώριο της ανάγκης. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο το πέμπτο τμήμα είναι ήδη στο περιθώριο έκθετη ανάγκη. Μία φορά μπορούμε να το δαπανίσουμε. Δεν μπορούμε να το δαπανίσουμε πολλέ φορέ, Πολύ απλά δεν γίνεται αυτό. Απευθύνω λοιπόν μια σαφή έκκληση προ του συναδέλφου. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε τη γερμανική και την ιταλική κυβέρνηση και το λέω αυτό γιατί ε, οι συνάδελφοι που είναι εδώ ήταν στην κυβέρνηση. Αυτοί μα έφεραν στο 12 μόριο γιατί δεν ήταν διτεθειμένοι να αποδεχτούν τον προϋπολογισμό αυτό θυσία. Και σε κάποιες περιπτώσεις ε, μιλάω και σε συναδέλφους που είναι από τα ίδια κόμματα που είναι στην κυβέρνηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίπτωση για την εισηγήτρια, γιατί είσαστε από το ίδιο κόμμα που κυβερνάει. Που έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα περάσουν όλα αυτά. Ούτε συζήτηση. Αυτό το λέω ξεκάθαρα γιατί δυσκολεύομαι λίγο. Θέλω πραγματικά να πετύχω μία πρόοδο να πετύχουμε. Και να επενθυμίσω και στο Γιάννου το εξή. Το 15-3 σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα έχουμε 300 εκατομμύρια επιπλέον. Σήμερα, μάλλον φέτος, μπορούμε να ζητήσουμε κάτι άλλο, το οποίο δεν πρόκειται να το πάρουμε. Αλλά το 15-3 σημαίνει 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο που θα έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιμένω και η προτεραιότητά μου είναι τα σημεία εκείνα στα οποία μπορούμε διαρκώς να έχουμε κάποια διαφορά. Εγώ βαστάω ως εισηγήτρια. Αλλά το τελευταίο πράγμα σας παρακαλώ πριν με διακόψει ο πρόεδρος ε, δικαίως και όλα γιατί μακρηγορώ. Ζητώ να καταλάβετε το εξής, ότι αν δεν αφήσουμε τα 900 εκατομμύρια την προηγούμενη φορά για ε, τους πρόσφυγες, σε μία στιγμή αναγκαστήκαμε να βρούμε ένα δις. Αν δεν έχουμε κάποιο περιθώριο, από πού θα το βγάλουμε αυτό το καινούργιο δισεκατομμύριο. Και αν πέρα από το δισεκατομμύριο παρουσιαστούν και κάποιες καταστροφές, τι θα κάνουμε. Η υπευθυνότητα σημαίνει ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι μέσα σε μία χρονιά μπορεί να παρουσιαστούν τέτοια έξοδα ύψου ενό δι και δεν θα έχουμε με τι να τα χρηματοδοτήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα ε, τη 30 Σεπτεμβρίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Α περάσουμε στο σημείο 9 της σα διάταξη, ενταλλαγή απόψεων σχετικά με την κτηριακή πολιτική των θεσμικών οργάνων. Κάθε χρόνο τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποβάλουν μια έκθεση όσον αφορά την κτηριακή του πολιτική στην αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή. Η προβλεπόμενη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων αποτελεί μια ευκαιρία για μα να καταλάβουμε καλύτερα την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, κτηριακή τη πολιτική τον Οκτώβριο θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την κτηριακή πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μωριό, ο οποίο είναι επικεφαλή τη Υπηρεσία Γραφείων και Υποδομών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Βρυξέλλε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε το λόγο. Έχουμε προετοιμάσει και μια παρουσίαση κύριε Πρόεδρε για το ζήτημα αυτό. και θα προσπαθήσω εν συντομία να σας, παρουσιάσω, την κτηριακή πολιτική που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Δεν λειτουργεί πολύ καλά από ό,τι φαίνεται το σύστημα. Μάλιστα. Πολύ σύντομα κάποια αριθμητικά δεδομένα. Το IOB διαχειρίζεται 61 κτίρια περίπου 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα ακαθάριστη έκταση, όπου έχουμε συνειδριακά κέντρα, διάφορες υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών και το καθεξής. Έχουμε λοιπόν περίπου 860.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Ένα μέρος της έκτασης αυτής χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως μας το ζητήσατε, σας παρουσιάζουμε εδώ πέρα ότι έχουμε 63% της επιφάνειας αυτής γραφείων ως ιδιόκτητα γραφεία και έχουμε και ένα 37% της επιφάνειας αυτής που είναι μισθωμένη επιφάνεια γραφείων, βραχυπρόθεσμα μάλιστα. Τα γραφεία αυτά βρίσκονται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Συνοικία αλλά και στον Πολιό και στη Γενέβη και έχουμε κοντά στην πλατεία Γοζιέ και κάποια γραφεία, ένα κτηριακό συγκρότημα που έχουμε κυρίως εκτελεστικούς ε, οργανισμούς. Ήδη από το 2007, στα πλαίσια της κτηριακής μας πολιτικής, έχουμε μία σταθερή γραμμή, η οποία έχει τους εξής τέσσερις άξονες. Πρώτον, επέκταση των ε, μισθώσεων, των ενοικηριστήριων συμβολέων, που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ο δεύτερος άξονας είναι η ανακαίνιση, η αναδιάρθρωση, η ανακατασκευή κάποιων ε, κτηρίων ιδιόκτητων που έχουμε, γιατί θεωρούμε ότι ε, τα κτίρια αυτά πρέπει προφανώς να πληρούν πάντα συγκεκριμένα πρότυπα, να έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο και γιατί ε, μπορούμε ενδεχομένω να θέλουμε να επεκτείνουμε μερικές φορές και τα γραφεία αυτά. Προχωράει πολύ γρήγορα. Βέβαια πρέπει ανατακτικά χρονικά διαστήματα να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η αγορά κινήτων, να γνωρίζουμε πώς έχει η αγορά αυτή, προκειμένου να ξέρουμε ποιες θα είναι οι μελλοντικές εξελίξεις και ποιες θα είναι οι μελλοντικές τιμές. Και βαθμία προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις λεγόμενες, τους λεγόμενους συνεργατικού χώρους εργασίας, να συστεγαζόμαστε ουσιαστικά με άλλες υπηρεσίες και άλλα γραφεία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο πλάζ. Το πλάζ είναι το τοπικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή διαχείριση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ισχύει επί του παρόντος. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν βελγικό νόμο που εγκρίθηκε πρόσφατα και ο οποίος απαιτεί μια μείωση της τάξης του 10% όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για τα επόμενα χρόνια με χρονικό ορίζοντα το 2025. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί σίγουρα θα επηρεάσει την κτηριακή μας πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Εντάχει, ποια είναι τα βασικά σημεία αναφοράς, αν θέλετε, της πολιτικής μας. Έχουμε το πλάζ, το πρόγραμμα αυτό το ανέφερα. Έχουμε έπειτα ήδη από τις αρχές του 2018 μια ευρεία έρευνα της αγοράς που κάναμε προκειμένου να δούμε ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για μας στο Μπολιό. Προτιμάζουμε τώρα μια βραχυπρόθεσμη επέκταση των γραφείων που έχουμε εκεί και έχουμε και κάποια μεγάλα έργα τα οποία προβλέπονται όσον αφορά για παράδειγμα την ανακατασκευή των γραφείων μας στην Rue de la Loi νούμερο 130. Εδώ πέρα η οικοδομική νομοθεσία που υπάρχει στο Βέλγιο μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον υπέργειο χώρο των γραφείων αυτών κατά 90.000 τετραγωνικά μέτρα και προβλέπεται και ένα νέο συνδριακό κέντρο 20.000 τετραγωνικών μέτρων το οποίο θα αντικαταστήσει το συνδριακό κέντρο Albert Borsette. Τώρα, όσον αφορά το κτίριο που βρίσκεται στην de la Loire, αριθμός 130, θα διαβάσετε σχετικές πληροφορίες και στον τύπο. τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα γραφεία αυτά. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο ρυθμιστικό γενικό σχέδιο, το οποίο προβλέπεται για την Ευρωπαϊκή Συνοικία για το 2008 και έπειτα έχουμε και τον σχετικό νόμο του Βελγίου όσον αφορά την κατασκευή στις αστικές περιοχές, νόμος του 2009 και έπειτα έχουμε και κάποιες εξαγορές κτηρίων για τις οποίες ενημερώσαμε την ε, αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή, όπως για παράδειγμα την αγοράσαμε το κτίριο Λουά 102 το 2016. Υπάρχουν λοιπόν κτίρια τα οποία ήδη μας ανήκουν, άλλα κτίρια τα οποία τα μισθώνουμε και υπάρχουν κτίρια τα οποία σχεδιάζουμε να αγοράσουμε τα ερχόμενα έτη. Επίσης, ξεκίνησε ένας διεθνής ερτεκτονικός διαγωνισμός τον Μάρτιο του 2018. Το Κολέγιο των Επιτρόπων πήρε την τελική του απόφαση τον Ιούλιο του 2019 και αυτή τη στιγμή προβλέπεται μια δημόσια έκθεση, είναι σε εξέλιξη ουσιαστικά, στο Γομπαν Σουμάν, στο ίνφοπόν που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ποιο κέρδισε το διαγωνισμό αυτόν. Ενδεχομένω το διαβάσετε στον τοπικό τύπο. Είναι διάφορα τα αρχιτεκτονικά γραφεία που συμμετέχουν στην αρχιτεκτονική αυτή κοινοπραξία. Έχουμε ένα ισπανικό αρχιτεκτονικό γραφείο που συνεργάζεται με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο βρετανικό και με ένα γερμανικό γραφείο αρχιτεκτόνων. Εδώ πέρα έχετε αρκετές λεπτομέρειες ενδεχομένως, πάντως σας περιγράφουμε πώς θα κινηθεί το όλο αυτό σχέδιο από τώρα μέχρι το 2025, ακόμα και 2030, όπου θα πρέπει να περάσουμε από διάφορα στάδια, ενημέρωσης επίσης της αρμόδιας για τον προπολογισμό αρχής. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την, το στάδιο εκείνο που προβλέπει διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο του διαγωνισμού αυτού όσον αφορά την πραγματική κατασκευή, την υλοποίηση του κυρίου αυτού. Να σας μιλήσω έπειτα για το νέο συνεδριακό κέντρο, ένα σχέδιο το οποίο φέρει τον τίτλο CC2.0. Εδώ πέρα έχουμε το κτίριο Αλμπέρα Μπορσέτα, κτίριο το οποίο είναι ιδιαίτερα παλαιό, μας προκαλεί πολλές δυσκολίες από τεχνικής πλευράς καταρχάς, γιατί θα πρέπει να συντηρούμε ανατακτικά χρονικά διαστήματα το κτίριο αυτό, προκειμένου να παραμένει επιχειρησιακό. Το κτίριο αυτό επίσης δεν αποκρίνεται πλέον στις ανάγκες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τρίτον, δεν έχουμε στο λεγόμενο αυτό συνεδριακό κέντρο τους απαραίτητου χώρους για να έχουμε πραγματικά συνέδρια. Μόνο κάποιες μικρές συνεδριάσεις τελικά μπορούν να γίνουν εκεί. Επίσης, Επίσης δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε πλήρως το κτίριο αυτό το οποίο το χρησιμοποιούμε ακόμα, επομένως μας δόθηκε η δυνατότητα να αγοράσουμε ένα νέο σύγχρονο κτίριο στην Ευρωπαϊκή Συνοικία. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε αυτό το οποίο ονομάζουμε ανταγωνιστικό διάλογο. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2017 υποβλήθηκαν κάποιε προφορέ, προσφορέ, τι οποίε αξιολογήσαμε μέχρι τον Ιούλιο του 2019 και αυτή τη στιγμή μα έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σχετική διαδικασία, δεν μπορώ να σα δείξω Εικόνε και φωτογραφίε από το τελικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Πάντω, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την ε, προσφορά αυτή που μα έχει γίνει και την οποία θα υποβάλουμε επίσημα στην αρμόδια δημοσιονομική αρχή μέχρι το τέλο του έτου. Και βέβαια χρειάστηκε να υπογράψουμε κάποιες ε, συμβάσεις και ελπίζουμε ότι η κατασκευή θα ολοκληρωθεί το 2023. Θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αφήσουμε το συνδρακό κέντρο Αλμπερ Μποσέτ και να πάμε στο νέο αυτό κτίριο. Τώρα, κάποιες ακόμα πληροφορίες ε, που καταδεικνύουν ότι τα θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Κάναμε μια ανταλλαγή κτηρίων με τις δύο επιτροπές, την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΕΟΚΕ. Έχουμε το κτίριο Βαν Μαντερλένα 2, το οποίο χρησιμοποιεί κυρίως η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία προτιμά να μείνει στο κτίριο αυτό, από το να μετατρέψει το κτίριο αυτό έπειτα σε γραφεία. Συμφωνήσαμε λοιπόν σε συνεργασία με την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών να κάνουμε μια ανταλλαγή κτιρίων, παίρνοντα εμεί δύο δικά του κτίρια και κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε και όλη αυτή τη διαδικασία κατεδάφιση, κατασκευή νέων κτηρίων και το καθεξής. Και μπορούμε επίση να διατηρήσουμε και τη γέφυρα αυτή που είναι υπέρια, που περνάει πάνω από την Γουλμπελιάχ και που επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στα κτίρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κτίρια τη ΕΟΚΕ και τη Επιτροπή των Περιφερειών. Πιστεύω ότι μέχρι το 2022 θα καταφέρουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις ανταλλαγές αυτές. Λοιπόν, έγινε η ανταλλαγή αυτή των κτηρίων, το κτίριο που βρίσκεται στην Πελιάρ 68 και το κτίριο που βρίσκεται στην Οδό Τχევ 74 και στις 28 Αυγούστου 2019 υπεγράφει η επίσημη συμφωνία ανταλλαγή των κτηρίων αυτών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δύο επιτροπών, Επιτροπή των Περιφερειών και ΕΟΚΕ δηλαδή. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο Akers Beckett από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ να σας αντιρρήσετε χρονικά όρια. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Να σας παρουσιάσω λοιπόν την πολιτική για την Λουξεμβούργο σε ό,τι αφορά τα πάρκινγκ. Βλέπετε λοιπόν τα τέσσερα κέντρα που έχουμε τα κτηριά μας ε, στο άνω τμήμα δεξιά. Έχετε το Κίσμπερκ, ιστορικά κτίρια της Κομισιόν στο Λουξεμβούργο. Έχουμε κάποια κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, το κτίριο ε, και και επίσης έχουμε το Ζαμονέ και κάποια προσωρινά κτίρια στο Κλώστορ, επίσης ε, κοντά στο Λουξεμβούργο και ένα κτίριο μια α, εγκατάσταση για φύλαξη κοντά στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Έχουμε λοιπόν περίπου 4.700 άτομα προσωπικό και 17 κτίρια. Τα πιο πολλά κτίρια είναι ενοικιαζόμενα με κάποιες ε, εξαιρέσεις όπου μπορούμε να αγοράσουμε τα κτίρια και αυτό μπορεί να αλλάξει λοιπόν στο μέλλον τα μεγάλα έργα τα οποία μας απασχολούν στην παρούσα φάση είναι το Ζαν 2, το μελλοντικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο που θα αντικαταστήσει το πρώην Ζαν Μονέ, το οποίο ουσιαστικά το έχει καταδαφίσει ο ιδιοκτήτης. Βλέπετε λοιπόν εδώ μία αρχιτεκτονική απεικόνηση του κτιρίου. Τρία κτίρια περιλαμβάνει, το χαμηλό κτίριο για 2.500 άτομα περίπου και ένα κέντρο συνεδρίων και εστιατόριο και ένα κτίριο, ένα πύργο που θα συμπεριλάβει ουσιαστικά γραφεία και ένα κέντρο υποδοχής. Και εγκαταστάσεις ασφαλείας για τους επισκέπτες ε, για όλα τα κτίρια, για τις ε, διασκέψεις. Οι εργασίες θα ξεκινήσαν μάλλον το Μάρτιο φέτο, φετινού έτους. Και μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες και πάλι. Μίλησα λοιπόν για τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα έργα αυτά. Τα βλέπετε στην διαφάνεια αυτή. Θα έχουμε λοιπόν περίπου 110.000 τετραγωνικά μέτρα στα κτίρια αυτά για 3.700 υπαλλήλου που θα μας επιτρέψουν ουσιαστικά να αφήσουμε όλα τα κτίρια τα οποία έχουμε στο Κλωστόχ. Και στο Κρυχμπερ και στο κέντρο. Εδώ πέρα βλέπετε και κάποιες ε, μακέτες και απεικονίσεις ψηφιακές των μελλοντικών ε, κτίριων, το auditorium, και επίσης στην καντίνα. Να σας πω τώρα τα υπόλοιπα έργα τα οποία θα θέλαμε να σας επισημάνουμε. Ποια είναι σε ό,τι αφορά την παράδοση του Ζαλμονε 2. Θα γίνει σε δύο φάσεις. Θα γίνει καταρχάς τον Φεβρουάριο του 2023 και το Φεβρουάριο του 2024 στη δεύτερη φάση. Έχουμε εναρμονίσει λοιπόν τα ενίκια των κτηριών, των προσωρινών κτηρίων, προκειμένου να είναι πιο ιδανικέ οι συνθήκε και να μην μείνουν άτυπα που να τα πληρώνουμε μέχρι τα, την παράδοση των ε, νέων κτηρίων. Θα σας στείλουμε επίσης ε, σχετικά σημειώματα ανακοίνωση για την ε, αντικατάσταση κτηρίων σε ό,τι αφορά πατικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις φύλαξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Σχολείων και θα είμαι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Κέλλερ. Στην κυρία Άγε, η οποία αντικαθιστεί την κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω τον κύριο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξήγηση αυτή να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της κυρίας Κέλλερ, η οποία μου ζήτησε να την εγκαταστήσω σήμερα. Κάνει πραγματικά πάρα πολύ προσεκτική δουλειά και ε, εξετάζει την κτηριακή πολιτική. Ήθελα λοιπόν να σας απευθύνω κάποιες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά και τα έγγραφα τα οποία είχε στη διάθεσή της για την προετοιμασία της παρουσίασης αυτής. Καταρχάς, στην παρουσίαση μιλήσατε για την ενεργειακή διαχείριση των κτηρίων στις Βρυξέλλες, αλλά δεν μιλάτε για την ενεργειακή απόδοση στο σημείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε σε ό,τι αφορά τη γενική πολιτική αυτή. Στο άρθρο 66 δεν ισχύει φυσικά, αλλά το New Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτάσσει να μειωθούν ε, οι εκπομπέ ε, διεξουδίου του άνθρακα σε ό,τι αφορά τα κτίρια. Δύο Δεν θα ήταν λοιπόν δυνατόν να ενταχθεί στο πλαίσιο των ε, αναφορών αυτών και η πτυχή αυτή και επίσης να μας μιλάτε για την βιωσιμότητα των κτίριων αυτών τι κόστος ε, ενεργειακό θα έχει η εκμετάλλευση των κτηρίων αυτών και ποιο είναι το κόστος ε, ανακαίνησης των κτηρίων. Μία άλλη ερώτηση σε ό,τι αφορά το πολιτές πρόγραμμα για την ε, μεταρρύθμιση των γραφείων, αναδιαρρύθμιση των γιατριών. Αναφέρεται απλά ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα μας διαβιβαστούν. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν. Πόσο έχει προχωρήσει λοιπόν το θέμα αυτό που θα μπορούσατε επίσης να μας δώσετε πιο πολλά στοιχεία για την αναθεώρηση αυτή και πότε θα γίνει η εγκατάσταση της Επιτροπής στα νέα αυτά γραφεία και θα έχουμε υπολογίσει τις νέες ε, ανάγκες. Επίσης, το, ε, ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Παρίσι από το 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το εγκατέλειψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλη 2018, γιατί το Συμβούλιο αποφανθήκε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή, ακριβό το εγχείρημα. Θα πρέπει να βρεθούν λοιπόν νέες εγκαταστάσεις για να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο και το καθεξής. Πρόκειται λοιπόν για ένα διαθεσμικό έργο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο, το οποίο προωθεί και τις εργασίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως στη σχετική έκθεση δεν αναφέρει τέτοια στοιχεία για το κτίριο αυτό. Θα πρέπει να προωθούνται αυτά τα διαθεσμικά έργα αλλά η συνεργασία αυτή δεν μπορεί να προκαλεί προβλήματα. Με ποια μέθοδο λοιπόν σκοπεύετε να... Με ποια μέθοδο σκοπεύετε να αποφύγετε τέτοια προβλήματα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στους σκιώδες η κυρία Χολμάιερ. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Και εγώ θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις για την ε, στρατηγική βιωσιμότητα. Υπάρχει τέτοια στρατηγική. Θα θέλαμε λοιπόν γραπτά να έχουμε στοιχεία για το ποια θα είναι τα σημεία προτεραιότητα και το πώ διαμορφώνονται τα πρότυπα ακριβώ, δηλαδή πώ εντάσσονται όλα αυτά στην κτηριακή πολιτική. Αυτά θα ήθελα λοιπόν να τα έχουμε γραπτά μπροστά μα και να αναφέρετε τα στοιχεία και οι προτεραιότητε και πώ εφαρμόζονται στην κτηριακή πολιτική. Κατά δεύτερον, αναφέρθηκε ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας στην, ε, στο Παρίσι. Και το κοινοβούλιο δεν έχουν νόημα τα κτίρια τα οποία είναι κάπου κρυμμένα σε κάποια γωνία και δεν περνάει ο κόσμος να τα δει. Αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει νόημα για διοικητικού σκοπούς, αλλά μα, για το Κοινοβούλιο χρειάζεται μεγάλη προβολή. Προκλήθηκε μεγάλη με μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά ένα κτίριο στη Βουλγαρία που έπρεπε κανείς να περάσει ε, από διεκπαιρεώσεις γιατί ήταν πίσω από μια προσβία το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι να είμαστε κάπου εμφανείς, να μας βλέπει ο κόσμος, όσο πιο πολλοί κόσμος γίνεται, να μπαίνουν ε, στην, ε, στα κτίρια μας, όχι να τα ξέρουν μόνο κάποιοι ειδικοί και εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς σκοπεύετε να ξαναξεκινήσετε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, ε, στην πλατεία Σούμαν υπήρχε με ένα σχέδιο για την ανεμόρφωση τη πλατεία. Τι γίνεται με αυτό, και τι σχέδια έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αγοράσει κάποια κτίρια τα οποία στο το παρόν εκμισθών και κάτι άλλο για το Λουξεμβούργο. Υπάρχει από πλευρά επιμελητία κάτι καλύτερο να μα προτείνετε σε σχέση με την δεκαετία του 80 για πρακτικούς σκοπούς. Ευχαριστώ κύριε Σουζακόφς. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Είμαι και εγώ νέο μέλος και χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω ακριβώ το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Κάποιες ερωτήσεις επιμέρους. Μπορείτε να μας δώσετε ε, στοιχεία για τα γραφεία στη Ρώμη, στο Δουβλίνο και στη Στοκχόλμη. Ε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι συμβάσεις ενοικίασης που έχετε φτάνουν στο τέλος τους. Ευχαριστώ κύριε Σαντρίσεν. Σας ευχαριστώ και για την έκθεση και για την παρουσίαση. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Η πρώτη ερώτηση. Την ακούσαμε στην παρουσίαση του κέντρου συνεδρίων που θα οικοδομηθεί το τωρινό κέντρο συνεδρίων. Χτίστηκε το 81, αν σωστά κατάλαβα. Ε, επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Μετά από 40 χρόνια ε, είναι μάλλον μία συνήθιση διάρκεια για ένα κτίριο. Τα 40 χρόνια. Δεύτερη ερώτηση αυτό το έγγραφο εργασία για το σχέδιο Γενικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 7ο τμήμα. Για αυτό το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη σελίδα 22 βλέπουμε μία σύνθεση για τα διάφορα κτίρια τα οποία είναι στο εξωτερικό και χρησιμοποιούνται ως αντιπροσωπείες διαπίστωσα ότι δεν έχουμε κανένα κτίριο στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Αυτό τι είναι, προσωρινό βήμα προκαταλαμβάνοντας το Brexit. Απλά μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η απάντηση. Τρίτη ερώτηση. Υπάρχει μήπως κάποιο κάποιος πίνακας για τις συντομογραφίες, για όλα αυτά τα κτίρια, γιατί δεν καταλαβαίνω ποια κτίρια είναι αυτά, δεν ξέρω καν πού είναι, πώς τα λένε και πού βρίσκονται. G12, G6, J16, υπάρχει κάπου ένας πίνακας για να βγάλω μία άκρη. Ευχαριστώ. Hm? Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα, λέει ο κ. Κούκς. John, you want to take the floor? So, uh, anybody else? Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο για τα κτίρια. Όχι λοιπόν. Ο κύριος Μουλινιό πρώτος και μετά ο κύριος Μπέκερ να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις γιατί το ΟΙΝΤΕ είναι κάτι το οποίο ανήκει ή μάλλον ασχολείται με ό,τι υπάρχει στις Βεξέλλες σε επίπεδο υποδομών και όχι εκτός βεξελων. Καταρχάς, καταλαβαίνω την ερώτησή σας για το ενεργειακό κομμάτι. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ακριβώς έθεσα το πρόγραμμα Plage το λαμβάνουμε υπόψη μας σε καθημερινή βάση. Η ενεργειακή αποδοτικότητα για τα παλαιά κτίρια δεν είναι αυτή που θέλαμε. Έχουμε κάνει προσπάθειες για να βελτιώσουμε τη μόνωση και τον κλιματισμό. Σεβόμεθα την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 3% κατέτος αλλά αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα επιπλέον πρέπει να περάσουμε σε νέα κτίρια. Και γι' αυτό ακριβώς ε, ξεκινάμε την υπόθεση ΛΟΑ 130, γιατί αν ε, μείνουμε ε, στα παλαιά κτίρια φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σωστά αποτελέσματα και δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τα υλικά τα οποία οδηγούν στη μείωση κατανάλωσης. Για το ΛΟΑ 130, αν δείτε τις δυνατότητες οι οποίες περιγράφονται στην προκήρυξη, πέρα από το ότι θα έχουμε ένα μέσο κατάλληλο για τους υπαλλήλους μας, λαμβάνουμε υπόψη μας κυρίαρχα τους περιβαλλοντικούς στόχους. Νομίζω επίσης ότι δεν είναι απίθανο να υπάρξει μια αναλυτικότερη παρουσίαση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έτσι και αλλιώς ο βελγικός νόμος μας υποχρεώνει, μας υποχρεώνει να παρουσιάζουμε μια έκθεση για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα πλαίσια της αιτήσιας, σε αιτήσια βάση Τώρα, τα στοιχεία τα οποία ακούστηκαν για το νίκο της Ευρώπης. Είναι κάτι για το οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, όμως η Γενική Διεύθυνση μας έχει ζητήσει βοήθεια σε επίπεδο συμβουλών ε, μηχανολόγους, μηχανικούς αρχιτέκτονες και διαχείριση προγραμμάτων έτσι ώστε κάποιες πιθανές αλλαγές στον τομέα αυτό να υποστηριχθούν από ειδικού που έχουμε εμεί στην υπηρεσία μας. Η βοήθεια αυτή ε, έγινε αντικείμενο μιας κάποιας συμφωνίας και θα στηρίξουμε την ε, γενική αυτή διεύθυνση σε τεχνικό επίπεδο. Σε τεχνικό, όχι σε πολιτικό. Τώρα για την ε, διάρκεια ζωής των κτηρίων. Εγώ καταλαβαίνω την, ε, την ερώτηση που εκπλήσεται για την σύντομη ζωή των κτηρίων είναι ένας από τους λόγους που μας κάνει να πούμε ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα το ΛΟΑ 130 έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε ένα κτίριο το οποίο να έχει ε, μία διάρκεια ζωής 2 επί 30 γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να, υπάρξει 60, 6, να υπάρξουν 60 χρόνια ζωής σε ένα κτίριο στο οποίο δεν θα παρέμβουμε και δεν θα σεβαστούμε τους νέους κανονισμούς για τα θέματα της ενέργειας. Συνεπώς, δυστυχώς, το CCAB ε, είναι ένα κέντρο το οποίο δεν ελέγξαμε στην κατασκευή του και εκείνη την εποχή κατασκευάστηκε με τον τρόπο αυτό και δεν προβλέπεται, επειδή ήμασταν και λίγα κρατημέλη εκείνα την εποχή, δεν προβλέπεται ένα συγκεκριμένος τρόπος για την ανακαίνισή του δεν μας παρέχει την ευελιξία την οποία θα επιθυμούσαμε. Πάντως είναι σαφές ότι στο μέλλον θέλουμε να αποφύγουμε. Τώρα για το Γενέβη 12 δεν καταλαβαίνετε βέβαια τα ονόματα και είναι λογικό και θα πρέπει να βάλουμε και τις διευθύνσεις ακριβώς για να μπορείτε να τα εντοπίζετε όλα αυτά στα έγγραφα τα οποία θα αναγνώσετε. Τώρα για το planning. Το πολιετές ε, πλαίσιο που είναι το γενικό πλαίσιο το οποίο αναπτύσσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κάνουμε για να έχουμε μία μακροπρόθεσμη εικόνα του τι ανάγκες θα υπάρχουν σε επίπεδο κτηρίων. Το ΛΟΑ 130 σαν παράδειγμα θα ξεκινήσουμε το 25 ένα πρώτο αποτέλεσμα το 30 και ένα δεύτερο το 35. Πρόκειται δηλαδή για σχέδια τα οποία είναι μακροπρόθεσμα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, ελπίζουμε πριν το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επομένου. Μιας και πρόκειται για ένα προγραμματισμό μακροπρόθεσμο και μιας και η πολιτική την οποία ακολουθούμε είναι σταθερή θα έλεγα, με τις ίδιες έννοιες δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις. Το planning λοιπόν το οποίο ακολουθείται στην παρούσα φάση είναι μια καλή αναφορά νομίζω σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπουμε στο μέλλον. Θα υπάρχουν ίσως κάποιες μικρές λεπτομέρειες, ίσως κάποιες μικρές παρατάσεις, αλλά μιας και οι εξελίξεις οι κατασκευαστικές δεν είναι πάντα οι επιθυμητές, παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσουμε. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις στις οποίες μπορούσα να απαντήσω. Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία άπτονται της Γενικής Διεύθυνσης Κόμμα να συμπληρώσω αυτά τα οποία ακούστηκαν για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το Ζάμονε 2 θα είναι σε επίπεδο Brian's. Το μελλοντικό κτίριο, το κέντρο των δημοσιεύσεων, που κατασκευάστηκε εδώ και 25 χρόνια και που ανταποκρίνεται θα έλεγα σε καλό επίπεδο στις ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτό ισχύει για τα κτίρια του Λουξεμβούργου αλλά και για ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων των Βρυξελών που είναι του τύπου έμας. Έμας είναι εγγύηση σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής αλλά και ε, ποσότητας ε, κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής αποβλήτων. Για το κτίριο CDE 6 θα σας στείλω στοιχεία για το κτίριο αυτό, το οποίο θα έχει ιδιαίτερα ικανοποιητικές ενεργειακές αποδόσεις. Για την επιμελητία είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην κυρία Χόλμαϊερ. Κατανοήσαμε το μήνυμά της και εμείς θα προχωρήσουμε ε, σε επιμέρους ρυθμίσεις όταν χρησιμοποιήσουμε το ζώμο 2 που θα μειωθεί το αριθμός των κτηρίων και ε, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε συγκεντρωτικά στα πλαίσια του 21ου αιώνα. Υπήρξε μια ερώτηση για τα κτίρια του Δουβλίνου. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να δώσει μια απάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το Λονδίνο αν κατάλαβα καλά και γιατί δεν υπάρχει στο κείμενο εργασίας στη σελίδα 22. Μιας και το έγγραφο αυτό είναι το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει τον, ε, την πρόταση προϋπολογισμού του 20. Ε, έλογα μπορούμε να αναμένουμε, δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύσει πια σήμερα βέβαια, αλλά μπορούμε να αναμένουμε ότι το 2020 δεν θα υπάρχει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο Λονδίνο θα υπάρχει μια μικρή αντιπροσωπεία γιατί τότε η Μεγάλη Βρετανία δεν θα είναι μέλος. Αλλά θα ζητήσω τη γνώμη των ε, υπευθύνων και αν μου δώσουν διαφορετικά στοιχεία θα επανέλθω. Καλώς σας ευχαριστώ, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Κλείνουμε το σημείο 9. Ευχαριστώ τις παρουσιάσεις, για τις παρουσιάσεις. Το σημείο 10, πολιετές δημοσιονομικό, 21-27. Έχει ξαναρχίσει η δουλειά για το πολιετές δημοσιονομικό με την ε, ε, σύσταση μιας επιτροπής διαπραγμάτευσης. Στα πλαίσια και των αποφάσεων της 16, 16 Σεπτεμβρίου του Συμβουλίου ε, παρουσιάστηκε η διαπραγματευτική ομάδα στο Κοινοβούλιο, ενημερωθήκαμε από τους Υπουργούς και για τις προθέσεις ε, του Συμβουλίου να δημοσιεύσει ένα έγγραφο τον Οκτώβριο πριν τη συνάντηση κορυφής για θέματα όπως το παγκόσμιο επίπεδο και η ισορροπία του πολιετούς δημοσιονομικού. Ε, αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές θα αναθεωρήσουν το κοιτίο διαπραγμάτευσης όπως λέγεται και γι' αυτό θα ήθελα από τον κύριο Όλμπριχτ και μετά την κυρία Μάρκες να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως το είπατε κι εσείς, η ε, διαπραγματευτική ομάδα συστάθηκε και έχουμε μάλιστα τώρα και δύο συνεισηγητές από τη μία πλευρά για το δαπάνε στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και δύο συνεισηγητέ έπειτα για του ίδιου πόρου. Και ήρθαμε σε επαφή και με την Φιλανδική Προεδρία του Συμβουλίου για να προετοιμάσουμε μαζί του το σχέδιο του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα, οι συναντήσεις αυτές που όπως είπατε συνδέονται με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων κινήθηκαν ομαλά, δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Μας ενημέρωσε το Συμβούλιο για τη δική του την πλευρά. Προτιμάζουν τώρα το δικό τους πλαίσιο διαπραγματεύσεων και ενώπιον του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου του Συμβουλίου θα προετοιμάσουν το σχέδιο τοποθέτησή τους. Δεν ξέρουν ακόμα τι θα περιλαμβάνει και ελπίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει μια πολιτική απόφαση πριν το τέλος του έτους. Θα πρέπει βέβαια οι συνάδελφοι να γνωρίζουν ότι το Nego Box, αυτό το κοιτίο, το πλαίσιο διαπραγματεύσεων, είναι ουσιαστικά η εσωτερική μέθοδος που ακολουθεί το Συμβούλιο, προκειμένου να προετοιμάσει τη θέση του για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και για τις τομεακές δαπάνες. Η μέθοδος αυτή που ουσιαστικά συνδέει το πολιετές δημοστομικό πλαίσιο και τους τομεακούς κανονισμούς είναι μια μέθοδος που τελικά αναμειγνύει τον κανονισμό του πολιετούς δημοστομικού πλαισίου με τους κανονισμούς των τομεακών δαπανών. Το πρόβλημα λοιπόν που δημιουργείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι εμείς για τους τομεακούς κανονισμούς έχουμε πολλούς διαφορετικούς εισηγητέ από διάφορες εμπλεκόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το Συμβούλιο λοιπόν προτιμάζει κατά αυτόν τον τρόπο την εσωτερική του τοποθέτηση, αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή καταλήξουν σε συμφωνία, ποια συμφωνία μετά θα παρουσιάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς για την πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες αποφασίσαμε να υποβάλουμε ένα ψήφισμα. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή κάποιους επιβασμούς επί του κειμένου αυτού, το οποίο θα ολοκληρωθεί λογικά την επόμενη εβδομάδα, αλλά πρέπει να κινηθούμε, όπως βλέπετε, σχετικά γρήγορα. Το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να, στήσουμε, να στείλουμε με, με το ψήφισμα αυτό. Εν γέννη, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι να υπενθυμίσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Νοέμβριο ήδη του 2018 να στείλουμε ουσιαστικά ένα μήνυμα στο Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει στην αρχική του τοποθέτηση που έγινε δεκτή από όλες σχεδόν τις πολιτικές ομάδες τον Νοέμβριο του 2018 και λέμε ουσιαστικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει στη θέση του αυτή. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει αν υπάρξει κάτι νέο στην πρόταση του Συμβουλίου, τότε αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται, να αντιστοιχεί μάλλον σε νέους πόρους, δηλαδή αν προβλεφθούν κάποια νέα καθήκοντα, οποιοδήποτε νέο καθήκον για παράδειγμα θα πρέπει να αντιστοιχεί και σε κάποια νέα χρηματοδότηση και κάτι άλλο το οποίο ζητάμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αν τελικά δεν υπάρξει συμφωνία έγκαιρη για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πριν τα τέλη του 2020 να προβλέπετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Είναι σε εξέλιξη όλη η εργασία όπως σας είπα. Αυτό που αποφασίσαμε στη χθεσινή μας συνεδρίαση είναι ότι ζητήσαμε ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει ήδη από τώρα να καταρτίζει το σχέδιο αυτό έκτακτη ανάγκης, προκειμένου να είναι διαθέσιμο αν προκύψει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση ή αν το Συμβούλιο δεν καταλήξει σε ομοφωνία ή αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά παρεμποδίσει την συμφωνία, αντιταχθεί ουσιαστικά στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Θα θέλαμε λοιπόν να καταρτήσουμε πολύ γρήγορα το ψήφισμα αυτό το οποίο θα έχει ένα έντονο πολιτικό χαρακτήρα στην πράξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει στην αρχική του θέση και αναμένει από το Συμβούλιο να καταλήξει στη δική του τοποθέτηση το συντομότερο δυνατό και λέμε επίσης ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ήδη από τώρα το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Βασικά το μήνυμα το οποίο αποστέλουμε στο Συμβούλιο είναι σαφέστατο. Λέμε ότι αν δεν λάβουν μια απόφαση μέχρι τα τέλη του έτους, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2020. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα θέλαμε εμείς να δείξουμε ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα plan B που εν προκειμένου θα είναι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Διάφοροι συνάδελφοι με ρωτούσαν σε ποιο βαθμό τελικά αυτή τη στιγμή πρόκειται να επαναλάβουμε το περιεχόμενο που είχαμε ήδη στην τοποθέτησή μας το 2018. Εμείς θέλαμε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ως προπολογισμό στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κάναμε και προτάσεις σε σχέση με συγκεκριμένε πολιτικές όπου πετούσαμε συγκεκριμένο προπολογισμό, συγκεκριμένα ποσά. Το θέμα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι να υποβάλουμε εκ νέου τα στοιχεία αυτά ή να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές βάσει των νέων προκλήσεων που καλούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε μεταξύ μας, γιατί έχοντας και πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γνωρίζουμε τώρα Μάλιστα εκπρόσωποι από τις επιμέρους γενικές διευθύνσεις μας ε, ενημέρωσαν ότι ε, ότι ε, πετύχαμε ουσιαστικά τον Νοέμβριο αντιστοιχεί σε ένα 25% χρηματοδότηση για τις δράσεις για το μετριασμό τη κλιματική αλλαγή στα πλαίσια του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα ενημερώνει ότι οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε πιο υψηλό ποσοστό χρηματοδότηση θα είναι κάπω προβληματικό. Εμεί πάντω εμένουμε στην αρχική μα τοποθέτηση. Είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε τι νέε αναδυόμενε προκλήσει, τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Πάντως είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσα σε δύο εβδομάδες να έχουμε εγκρίνει το ψήφισμά μας, το οποίο όπως σας είπα θα είναι έτοιμο το σχέδιο του κειμένου στο τέλος της επόμενης εβδομάδας και δεν θα έχουμε τις απαραίτητες βέβαια πληροφορίες για να μπούμε σε πολύ λεπτομεριακή ανάλυση όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα. Συνοψίζοντας λοιπόν, όσον αφορά τις δαπάνες, διατηρούμε την αρχική μας θέση, αυτή που εκφράσαμε δηλαδή τον Νοέμβριο του 2018. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει ήδη από τώρα να επεξεργάζεται το σχέδιο έκτατης ανάγκης και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να αναλύουμε την νέα αναδυόμενη κατάσταση Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι στο πλαίσιο του ψηφίσματος αυτού να μην αλλάξουμε την αρχική μας θέση, δηλαδή το 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος να δίδεται ως συνεισφορά από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα έχουμε λοιπόν το κείμενο έτοιμο, όπως σα είπα, μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας και αν πραγματικά θέλετε να εγκρίνουμε το κείμενο αυτό στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου, όλες οι σχετικές εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Εξού και ο επίγον χαρακτήρα του εγγράφου αυτού. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκέ, έχει το λόγο. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπε ο συνεισηγητής, όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή. Θα ήθελα απλώς και νομίζω ότι ήδη έκανε αυτή τη στιγμή μια σχετική ανάλυση ο προλαλής σας, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την αρχική τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια έκθεση, ένα κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντιστοιχεί στη θέση του και θα πρέπει ακριβώ αυτό να φαίνεται στο ψήφισμα αυτό το οποίο θα εγκρίνουμε. Τώρα, ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών δεν προέκυψαν ουσιαστικά κάποιες νέες προκλήσεις, απλώς Προσπαθήσαμε μέσω συγκεκριμένων πολιτικών να αποκριθούμε σε κάποιε έκτακτε καταστάσει οι οποίε προέκυψαν. Για παράδειγμα, έκτακτε καταστάσει που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματο στηρίζουμε την πρώτερη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση για την κλιματική δράση. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε κάποιες από τις αρχές που προέβαλε και η ίδια η νέα πρόεδρος Φοντερ Λάιλεν όσον αφορά την παρουσίαση ενός νέου εγγράφου από την Προεδρία. Εμείς ήδη τον Απρίλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβαμε την πρώτη ανακοίνωση καταλήξαμε σε, μία, συναψήφισμά ένα ψήφισμά μας το Νοέμβριο και η Προεδρία τώρα του Συμβουλίου από ό,τι φαίνεται θα παρουσιάσει ένα νέο έγγραφο αφού του ήρθε σε επαφή πρώτα με τα κράτη-μέλη αφού έκανε τις απαραίτητες διμερείς συναντήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι ε, δύο είναι εναλλακτικέ. Είτε θα υποβληθεί ένα νέο έγγραφο από την Προεδρία που θα βασίζεται στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις απαραίτητες προσαρμογές βέβαια που απορρέουν από τις διμερείς αυτές επαφές ή η Προεδρία θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό εναλλακτικό έγγραφο. Αν πραγματικά το Συμβούλιο θέλει να στείλει ένα μήνυμα διαλόγου όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει ουσιαστικά να καταφέρει να προσεγγίσει λίγο περισσότερο τη δική μας την τοποθέτηση που είναι ήδη γνωστή στο Συμβούλιο από τον Νοέμβριο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει το Συμβούλιο, αν πραγματικά θέλει να έρθει πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συμπεριλάβει στο κείμενό του κάποια από τα στοιχεία, κάποιε από τι προτάσει και τα αιτήματα που έχει παρουσιάσει το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, το σχέδιο έκτακτη ανάγκη στο ψήφισμά μας αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο να αποτελεί ένα plan B. Θέλουμε ένα σχέδιο το οποίο να ανταποκρίνεται στην κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Αν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία κατά τη διάρκεια του 2019, τότε θα πρέπει όντως να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου τα κράτη-μέλη, οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορέσουν να συνεχίσουν ομαλά και απρόσκοπτα να υποφελούνται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς να προβλέπετε κάποια διακοπή στη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα τους συνεισηγητές και τους εισηγητές για τους ιδίους πόρους. Η κυρία Αγία πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Φερνάντες, σα ευχαριστώ που μου δίνετε κατά προτεραιότητα το λόγο. Νομίζω ότι έχουμε κάθε συμφέρον να προχωρήσουμε με τέτοια ταχύτητα έτσι ώστε να ακουστούν οι ανησυχίες μας. Τρία σημεία. Πρώτον, να επιμείνω στο κατεπήγον του θέματος. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό. Είναι μια, υπάρχει μια ομάδα εδώ νέων βουλευτών, οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν φυσικά τα πράγματα και δεν ξέρουμε επί της ουσίας τη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό και τους ιδίους πόρους. Στόχος είναι να υπάρξει ένα μήνυμα, ένα ψήφισμα προς το Συμβούλιο ότι είμαστε έτοιμοι και είμαστε ενωμένοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο να μην ξανανοίξουμε την, το κουτί της Πανδώρας ΕΛΚ, ε, Σοσιαλιστές, Ρινιού και Πράσινοι. Για να μην γίνουν εκ νέου οι συζητήσεις οι οποίες είχαν προηγηθεί στο παρελθόν και οι, οποίοι οι οποίες θεωρήθηκαν όλο ότι ολοκληρώθηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Ζητάμε κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου και του φιλόδοξου προγράμματος ε, της Ουρσουλα Φοντερ Λάιεν σε αυτό αναφέρθηκε ήδη ο Γιάνν και η Μαργαρίτα. Ε, το θέμα το κλιματολογικό είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ομάδα μας. Ο Μωρίς ίσως να μιλήσει και για τα θέματα του κράτους δικαίου. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο εργασίας επί ενός κειμένου ε, ισχύρου, φιλοδόξου αλλά και συνενετικού για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή ακριβώς πλειοψηφία και δεν ξέρω αν ε, ο, Χωσέ, Ζωζέ Μανουέλ θέλει να πει κάτι πιο συγκεκριμένο για τους ιδίους πόρους. Ο κ. Φερναντές έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που έκαναν ο εισηγητής Γιάνν Όλμπριχτ, η κυρία Τομά, ο κύριος Λεβαντόφσκι και ο Ζεράρ Ντεπρέ, γιατί μας άφησαν θα έλεγα μια πολύ μα πολύ καλή κληρονομιά. Πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση και η οποία χαρακτηρίζεται και από την ορθή μεθοδολογία. Η μεθοδολογία την οποία ακολουθούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι όπως είπα η σωστή. Βλέπουμε τι χρειαζόμαστε για κάθε πολιτική και μετά κάνουμε την πρόσθεση. Από κάτω προς τα πάνω. Ενώ το Συμβούλιο ακολουθεί το αντίθετο. Το Συμβούλιο λέγει ότι βάζουμε ένα ανώτατο όριο και μετά κάνουμε κατανομές και διαιρέσεις. Και με το 1% προφανώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πολιτικές προκλήσεις. Ένας μικρημένος προϋπολογισμός είναι κάτι το πάρα πολύ κακό και οδηγεί στο να πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τελικά το μικρό προϋπολογισμό. Επιμένουμε φυσικά και στους νέους ιδίους πόρους. Ιδίους πόρους οι οποίοι φυσικά προασπίζουν ε, την δημοσιονομική ουδετερότητα που χρησιμεύουν στην χρηματοδότηση νέων πολιτικών. Αν πράγματι θέλουμε εμείς να μειώσουμε ε, τα χρήματα τα οποία δίδουν ε, τα κράτη-μέλη με βάση το ΑΕΠ, τότε θα πρέπει από την άλλη να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό και νομίζω ότι το 1,3 ΑΕΠ για τον προϋπολογισμό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θυμίζω αυτό το οποίο επανειλημμένα έχουμε πει, δεν θα υπάρξει συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Κοινοβούλιο για τους νέους ιδίους πόρους. Μια συμφωνία που σημαίνει νέους ιδίους πόρους, σημαίνει επίσης διαφάνεια, σημαίνει απλοποίηση, σωστούς μηχανισμούς αντιστάθμισης και ένας προϋπολογισμός διαφανής και αναγνώσιμος. Είμαστε έτοιμοι, είναι κατεπήγον το θέμα. Βλέπουμε ότι το Συμβούλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Δεν ξέρω αν η Προεδρία αυτή τη στιγμή κάνει ένα παιχνίδι για να μειώσει ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες που υπάρχουν αλλά η μείωση της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το χείριστο μήνυμα είναι το χείριστο μήνυμα γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν έχει νέες φιλοδοξίες και νέες φιλοδοξίες για μας σημαίνει νέες πράξεις, νέες φιλοδοξίες, νέες επιπλέον αυξήσεις, προσθέσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέες πολιτικές, για ενίσχυση των ισχυουσών πολιτικών, απαιτούνται νέα μέσα, οι πολίτες περιμένουν έναν προϋπολογισμό συνολικά σημαντικό, όλοι να ωφεληθούν και να καλύψουν τις ανάγκες αυτό το οποίο ζητά και το Κοινοβούλιο. Ενωμένο. Αντρέσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Ούλμπριχτ και τους προηγούμενους βουλευτές που πήραν τον λόγο και τους βουλευτές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου και βοήθησαν στο Κοινοβούλιο να προετοιμαστεί σωστά και να μπορέσει να διαπραγματευτεί σωστά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν εξ αρχής θα πρέπει να προσθέσουμε νέες προτεραιότητες για μας, για τους πρασίνους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ε, μια σωστή συζήτηση για το λεγόμενο Green Deal της Φόντερ Λάιεν, της Προέδρου. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο... Έχει μια πολύ καλή θέση και θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και σε ό,τι αφορά την, ε, τον εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά ε, τη χρηματοδότηση των μεγάλων μελλοντικών προκλήσεων. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να πω ξεκάθαρο το γεγονός ότι για παράδειγμα η γερμανική κυβέρνηση κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει τη, σε ό,τι αφορά του μεγάλου συνασπισμού και δηλώνει ότι δεν επιτίθεται να χρηματοδοτεί πλέον τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και νομίζω ότι εδώ είναι δικό μας καθήκον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τι εθνικές κυβερνήσεις γιατί τα κράτη-μέλη, τα μεγάλα, τα πλούσια κράτη-μέλη όπως η Γερμανία για παράδειγμα δεν μπορούν μόνο να εκφωνούν ωραίους λόγους σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα πρέπει συγκεκριμένα να καταδεικνύουν την υποστήριξή του όταν κάνουμε διαπραγματεύσει εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Και κυρίως η γερμανική κυβέρνηση έχει μεγάλο ρόλο και μεγάλη ευθύνη γιατί είναι τόσο μεγάλο κράτος μέλος η Γερμανία και κινείται προ τη λάθο κατεύθυνση. Θα πρέπει είτε να υπάρχει μεγαλύτερη ποσοστία συμμετοχή στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή να ε, δώσει τη δυνατότητα για την επιβολή ευρωπαϊκών φόρων. Και αυτό αποτελεί μια δυνατότητα. Θέλουμε λοιπόν έναν ανεξάρτητο και ισχυρό προπολογισμό και θα μπορούσε να υπάρχει λοιπόν και ψηφιακό φόρο, ένα φόρο διοξιδίου άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίο θα πηγαίνει κατευθείαν στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μέσω των εθνικών προπολογισμών. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε αντιτεθειμένοι να επενδύσουμε στο μέλλον μα, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε έτσι λύση και συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Φερνάνδες και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε ως απόψη μας προς το Συμβουλίο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουαλμίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως η εισηγήτρια για τους σοσιαλιστές ξεκινάω από το εξή. Κάτι που με ιδιαίτερα προσφυλές και το τόνισε και ο κύριος Φερνάνδε, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνδέσουμε τις διαπραγματεύσεις μας αυτές για τους ίδιους πόρους με τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο θέλουμε όσον αφορά την αναθεώρηση των ιδίων πόρων. Αυτό το πρώτο σημείο νομίζω ότι βρίσκει σύμφωνο και του υπόλοιπου συναδέλφου και για μένα είναι καθοριστική σημασία. Όσον αφορά τώρα τι προτινόμενε μεταρρυθμίσει για, για του ίδιου πόρου, τον Μάιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τέσσερα επιμέρου έγγραφα με τέσσερι προτάσει για τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων. Αποτελούν βάση για την έναρξη των συνομιλιών, θεωρώ. Αλλά όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, Νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι αυτή τη φορά. Ένας πρωταρχικός μας στόχος ε, είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το σύστημα των ιδίων πόρων λιγότερο ασαφές και πιο διαφανές. Να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι ποσοστώσεις ενισφοράς σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με ένα ακόμα στόχο που έχουμε, δηλαδή να μειώσουμε τα ποσοστά αυτά συνεισφοράς των κρατών μελών, προσθέτοντας όμως νέα τέλη, νέα έσοδα στους ιδίους πόρους, έστω τα οποία θα είναι καθαρά ευρωπαϊκής όμως φύσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει κάνει κάποιες σχετικές προτάσεις, για παράδειγμα η συνολική αυτή φορολογική βάση, μία, ένας φόρος που θα μπορούσε να έχει να κάνει με τις πολυεθνικές εταιρείες και που αν εφαρμοζόταν νομίζω ότι θα πετύχαινε και τους στόχους που έχουμε για την κοινωνική δικαιοσύνη και εν γέννη για την φορολογική ευθυγράμμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση του φόρου που προβλέπεται στα πλαίσια του συστήματος εμπορίας εκπομπών και εμείς μπορούμε να το δεχθούμε αυτό και προβλέπεται επίσης και ένας φόρος να τέλος για τα μη ανακυκλώμενα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίε. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας τις νέες αυτές προτάσεις, να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα τους ιδίους πόρους με καθαρά ευρωπαϊκές αν θέλετε πηγές και να μειώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο το, τη συνεισφορά των κρατών μελών. Και επίσης θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο και την ιδέα του ψηφιακού φόρου. Δηλαδή να έχουμε έναν φόρο όσον αφορά τις ψηφιακές συναλλαγές ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουμε το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή ακόμα και των μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν νέα έσοδα για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέους ιδίους πόρους και μπορούν να χρηματοδοτήσουν καλύτερα τον προπολογισμό έχοντας μια καλύτερη ανακατανομή των συνεισφορών που θα πρέπει να γίνουν προ τον κοινοτικό προπολογισμό, που θα πρέπει να γίνουν αυτή τη φορά και από τι πολυεθνικέ επιχειρήσει και από τι επιχειρήσει τη ψηφιακή τεχνολογία. Και νομίζω ότι υιοθετώντα επίση και τον φόρο αυτό για τον άνθρακα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και του στόχου τη κλιματική αλλαγή. Τέλο, δεν γνωρίζουμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση με το Brexit και εγώ ίδια ως πολιτολόγος δυσκολεύομαι ιδιαίτερα να καταλάβω τελικά τι μέλη γενέστε. Αν όντω αποχωρήσει πάντως το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να καταργήσουμε όλη αυτή την έκπτωση, την επιστροφή που προβλεπόταν στο πλαίσιο του ενωσιακού προπολογισμού που οδηγούσε σε τεράστιες αδικίες και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την εξηγήσουμε την έκπτωση αυτή προς τα έξω. Και επίσης δύσκολα γινόταν αποδεκτή από τα κράτη-μέλη στα βόρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα γίνει με μία ανακατανομή των πιστώσεων και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες άλλες πιστώσεις προκειμένου να αυξήσουμε τον κοινοτικό προπολογισμό. Καλύτερη κατανομή λοιπόν των πιστώσεων, απλούστευση του όλου συστήματος, καλύτερη χρησιμοποίηση άλλων τελών και εσόδων και μια απλούστευση του φορολογικού συστήματος στα κράτη-μέλη. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε πραγματικά έσοδα τα οποία να προκύπτουν από πραγματικές ευρωπαϊκές ενωσιακές πολιτικές. Ελπίζω να το πετύχουμε λοιπόν το στόχο αυτό και ελπίζω πραγματικά οι προσδοκίες μας αυτές να αποτελέσουν πραγματικά από το τμήμα των επερχόμενων διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κύριε Κολνέρα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ως κοιόδης εισηγητής για την ε, ομάδα Renew, έκανα πραγματικά πολλές έντονες συζητήσει με πολλούς βουλευτές για το Πουδουπού, γιατί προφανώς όλοι ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι είναι ισχυρή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επίσης θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την τοποθέτηση του προηγούμενου Κοινοβουλίου, θα πρέπει να αποτυπώσουμε τις προτεραιότητες της Νέας Επιτροπής και θα πρέπει να προωθήσουμε προκειμένου να μην ε, παραμεριστεί αυτό το σχέδιο, αυτό το σχέδιο ανάγκης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτό το ποδοπού να τονίσουμε την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Χρειαζόμαστε αύξηση του προπολογισμού. Θα πρέπει να πολεμήσουμε να το πετύχουμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, γιατί αυτή η ενέργεια, αυτές οι ενέργειες ε, αξίζουν πιο πολύ από ότι οι μεμονωμένε δράσει των μεμονωμένων κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να το δείξουμε αυτό και προ του πολίτε, ότι επενδύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση τελική ανάλυση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για την ε, ομάδα του Renew. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα μηχανισμό ε, κράτου δικαίου σε ό,τι αφορά τον πολιτευτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με τον τρόπο αυτό. Επίσης, σε ό,τι αφορά το... τη ρήτρα κράτου δικαίου, θα πρέπει να μείνουμε να μπει στον προπολογισμό και προσβλέπω πραγματικά στη μελλοντική μας συνεργασία. Θεωρώ ότι έχουμε μια σημαντική ευκαιρία για να καταρτήσουμε ένα σωστό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσάνη. Ε, Ευχαριστώ. Κάποιες ε, σκέψεις γενικού τύπου για, το, για την πορεία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα και για το τι ακολούθησε μετά τη διακοπή των ευρωπαϊκών εκλογών πάνω στα ένα από τα δύο θέματα τεστ με τα οποία θα ασχοληθεί η ευρωπαϊκή πολιτική. Ένα είναι το πολιετές και ένα άλλο είναι το Brexit, το οποίο θα επηρεάσει έτσι και αλλιώς το ε, πολιετές δημοσιονομικό. Τώρα για το χρονισμό. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Φιλανδική Προεδρία θέλει να κλείσει τη συζήτηση με μια συμφωνία πριν το τέλος της δικής της περίοδου, αλλά κατ' εμέ υπάρχουν σημαντικές διαιρέσεις και προβλήματα και στο εσωτερικό του Συμβουλίου και σε σχέση με αυτά τα οποία θέλουν τα κάνουν τα κράτη-μέλη. Ορισμένες χώρες θέλουν ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο, κάποιες άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να μειώσουν τους αριθμούς οι οποίοι προτείνονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο. Εγώ θυμίζω ότι για τα θέματα του χρονοδιαγράμματος ήδη το προηγούμενο Κοινοβούλιο και η προηγούμενη Επιτροπή είχαν προσπαθήσει να κλείσει πριν το τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου, κάτι το οποίο δεν έγινε. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθήσουμε τον χρόνο που έχουμε πλέον υποχρεωτικά ε, να τον εκμεταλλευτούμε και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω ρήγματα θεσμικά μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και σχετικά τώρα με το χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις, το κοινοβούλιο του, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έχει συνδέσει την σύνδεση με τους ιδίους πόρους με τη Γενικότερη Συμφωνία. Εγώ βλέποντας ε, τις πολύ μεγάλες δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν για να καταλήξουμε στον τομέα της, των ιδίων πόρων, ε, έχω την αίσθηση ότι το να βάζουμε από κοινού αυτές τις δύο διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο θα επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό. Οι δυσκολίες είναι διαφορετικές και το να τα βάλουμε όλα σε ένα πακέτο είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την συζήτηση για το πολιετές. Σχετικά τώρα με το περιεχόμενο των προτάσεων. Έχουν καθοριστεί ορισμένες νέου τύπου προτεραιότητες και τουλάχιστον στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αν θέλουμε όμως εμείς να χρηματοδοτήσουμε μια νέα, προτε... μια νέα αν θέλετε, προτεραιότητα, τότε θα πρέπει να ασχοληθούμε με πολιτικές οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη συνοχή μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές στο εσωτερικό της Ένωσης και την κοινή αγροτική πολιτική, ένα γεωργικό τομέα ο οποίος αντιμετωπίζει και για εσωτερικούς λόγους και για εξωτερικούς λόγους πολλά προβλήματα, σαν παράδειγμα κυρώσεις και αντικυρώσεις επηρεάζουν αρνητικά τον γεωργικό τομέα. Νομίζω λοιπόν ένας ρεαλιστικός τρόπος αντιμετώπισης που σέβεται τις ιστορικές προτεραιότητες είναι προτιμότερος και θα βοηθήσει τις επιδόσεις του προϋπολογισμού μας με θετικό τρόπο. Κλείνω με μια γρήγορη αναφορά στους ιδίους πόρους. Και εδώ ε, νομίζω ότι είναι απαραίτητος ο στόχος της μείωσης των πιστώσεων από πλευρά των κρατών μελών, χωρών όπως ε, η Ιταλία που είναι καθαρή συνεισφορής, εισφορής που έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει βέβαια εις βάρος, ή μάλλον μέσω της επιβολής νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και δεν θα πρέπει να έχει την δυνατότητα φορολόγησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος και οι προτάσεις οι οποίες ακούγονται ε, και από την ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ιδίους πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθούν μια κατεύθυνση η οποία στην ουσία μας οδηγούν στη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών και από την άλλη βάζουμε φόρους οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, φόροι οι οποίοι μπορεί να έχουν, ε, αν θέλετε, ε, να είναι ελκυστικοί σε επίπεδο μάρκετινγκ και διαφήμισης, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το τι θα ακολουθήσει στο πολιετές δημοσιονομικό. Ευχαριστώ. Τσίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, εξ ονόματος του ECR θα ήθελα να πω ότι δεν είμαστε μέλη τη Σώματο Εργασία, αλλά και εμεί θέλουμε να συμβάλλουμε για την κατάρτιση του πολιτικού δημοσιονομικού πλήσου σε ό,τι αφορά το σχέδιο ε, ανάγκη, το οποίο ανέφεραν οι συνεισηγητέ. Καταρχά, συμφωνούμε με την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το πουδουπού για τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τη τεχνική διάσταση. Δεν μπορούμε να πετύχουμε οποιαδήποτε συμφωνία για το που το που, αν δεν ε, βρούμε μια συμφωνία για τους ίδιους πόρους της Ένωσης. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε στα χέρια μας. Κατά δεύτερον, χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Συμφωνούμε με τον κύριο Ολμπρίχτ σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να καταλάβουμε επίσης και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε λοιπόν πιο πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τον προπολογισμό και πράγματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη σε ό,τι αφορά και τις δαπάνες ε, και τα έσοδα. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα ή άλλους επιπλέον πόρους που χρειάζονται. Επίσης, η άλλου επιπλεον πορου που χρειαζονται επισης η αιρεσιμοτητα για το κράτο δικαίου, που είναι αμφιλεγόμενο θέμα. Καταλαβαίνετε τη θέση μα ε, από πλευρά του ECR και αυτό λοιπόν συνδέεται με θέματα προπολογισμού Και εδώ πρέπει να κατανοήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ πέρα θα μπορούσαν να υπάρχουν και επιπλέον ήδη πόροι σε ό,τι αφορά τη φορολογήση του άνθρακα, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε τι ισχύει και για τρίτες χώρε όμω όπου εισάγουμε για παράδειγμα προϊόντα και είναι πολύ λιγότερο βιώσιμη η όρη στα ορίχια. Επί τη ουσία δύο κουμπέντε να πω, νομίζω ότι το ECR πάντα ήταν υπέρ τη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξίας και εδώ ιδιαίτερα στον τομέα τη αγορά και των υπηρεσιών είμαστε υπέρ τη ευρωπαϊκής διάστασης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις ανάγκες του Πουδουπού με τις προσδοκίες των πολιτών. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ε, εκ βάθρων, για παράδειγμα, θέματα ε, διευθυντικής πολιτικής. Το διευθυντικό ταμείο έχουν κάποιες ε, προσδοκίες οι πολίτες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και την πολιτική γεωργίες που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί κάποια στοιχεία και να δούμε και τα νέα τμήματα του που, που τα προγραμμάτα ορίζουν κτλ αυτές ε, οι μικρολεπτομέρειες οι οποίες όμως κάνουν διαφορά, ιδιαίτερα όταν η οικονομία είναι σε ύφεση. Η μακροοικονομία στην ε, Γερμανία και στην Ολλανδία έχει αλλάξει. Έχουν ε, διαθέσει να κάνουν μεγαλύτερε δαπάνε. Αλλά να δούμε τι γίνεται με τι σύμβολες βάσει του ΑΕΠ. Η πιο μικρή συνεισφορά θα σημαίνει και λιγότερη συμμετοχή στι διεθνεί αγορέ. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει τις διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι θα επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το 1,3% του ΑΕΠ. Εδώ θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το ποσοστό, αλλά να δούμε και που μπορούμε να κερδίσουμε πιο πολλά στοιχεία σε από πλευρά ποιότητα και ουσία. Ευχαριστώ, κύριε Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής ε, ε, περίοδου είχαμε εντελώς μη ρεαλιστικές ή αφελείς αν θέλετε προσδοκίες για το τι θα πετυχαίναμε για μετά τις εκλογές και είχα πει όντω τότε στους συναδέλφους ότι δεν ήταν ρεαλιστικές οι προσδοκίες μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ε, κατά τη διάρκεια της περίοδου των εκλογών τοποθετούμασταν όσον αφορά την ε, μετεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις είναι καθαρά διακυβερνητικές. Δεν έχει εμπλακεί τουλάχιστον ουσιαστικά ακόμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα γίνει μόνο όταν θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι ε, δύο τουλάχιστον συνεδριάς του Συμβουλίου και όχι μόνο μία απαιτούνται. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι στις αρχές του 2020 θα καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία και όχι στην πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου, εκτός και αν γίνει κανένα θαύμα, ποιος ξέρει. Μπορεί με τις εξελίξεις που θα έχουμε στο Brexit να καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία με την πρώτη απόπειρα που θα κάνουμε. Πάντω, σε κάθε περίπτωση νομίζω τελικά στι αρχέ του 2020 θα καταφέρουμε να έχουμε διαπραγματεύσει για τον βασικό κανονισμό. Θα ακολουθήσουν και άλλε διαπραγματεύσει όσον αφορά του τομεακού κανονισμού στη συνέχεια. Όσον αφορά του ιδίου πόρου. Το Brexit εδώ πέρα μας προσφέρει μια ευκαιρία. Θα θυμάστε κάποιες προτάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, οι οποίες δεν ευωδόθηκαν γιατί είχαμε τότε μία άτεγκτη στάση του Κάμερον απέναντι προτάσεις που έκανε η ομάδα του Μόντι. Τώρα θα μπορούσαμε να είχαμε κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις όσον αφορά την φορολογία των εταιριών ή το φόρο προστιθέμενης αξίας. Ίσως τέλος πάντων μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα των ιδίων πόρων. Το παράδοξο τώρα είναι ότι έχει επικριθεί τόσο πολύ το σύστημα αυτό ότι βρήθη τελικά εξαιρέσεων και ειδικών καταστάσεων, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει απαραίτητη πρόθεση μεταρρύθμισής του. Η κυρία Γκαρθιαμπάλ Ρουμπιάλ έχει το λόγο. Πράγματι θα πρέπει να εγκρίνει μία πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την οποία είχαμε ήδη ψηφίσει στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τον πιο σαφή τρόπο τους αριθμούς, τα ποσά και έτσι να επιτρέψουμε και στους νέους βουλευτές είναι κατανοηθό αυτό να μπορέσουν να ενσωματώσουν, να κατανοήσουν τις θέσεις τις οποίες θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Και σημασία έχει το Συμβούλιο να κατανοήσει ότι επιτέλους υπάρχει το Κοινοβούλιο Εμείς ήδη από το 18 έχουμε καταλήξει σε κάποιες θέσεις και προσπαθούμε να κατανοήσουμε ποια θα είναι η απόφαση και οι προτάσεις του Συμβουλίου. Και σε επίπεδο εσωτερικό και σε επίπεδο εξωτερικό λοιπόν έχουμε κάνει κάποιες ε, προτάσεις. Τώρα ε, πρώτον μιας και έχουμε μια νέα επιτροπή και με μια νέα πρόεδρο μπορούμε να καταλήξουμε σε νέους στόχους, σε νέες προτεραιότητες, σε νέες κοινέ προτάσεις και να επαρκεί ποσά για τη χρηματοδότηση όλων αυτών. Γνωρίζουμε επίσης ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο και δεν μπορούμε μετά από τόσα χρόνια διαπραγμάτευσης να μην καταλήξουν σε μια συμφωνία εμείς να πούμε ότι αυτή είναι η πρότασή μας και να πιέσουμε έτσι ώστε να γίνει δεκτή για πολιτικής όπως οι πολιτικές συνοχής και άλλες κοινοτικές πολιτικές. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει πια ιδιαίτερος χρόνος. Γνωρίζει το Συμβούλιο ακριβώς τις δημοσιονομικές συνέπειες των προτάσεών μας και γνωρίζει ότι εμείς δεν θα διστάσουμε να πούμε όχι αν τυχόν δεν υπάρξει συμφωνία για τους ίδιους πόρους. Λοιπόν, εμείς ξεκαθαρίσαμε τις προτεραιότητές μας, ξεκαθαρίσαμε ποιοι είναι οι στόχοι που έχουμε, επαρκείς ήδη οι πόροι βασικά, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα οποία αποφασίζουμε σε δημοσιονομικό πλαίσιο και καλό θα είναι επιτέλους το Συμβούλιο να καταφέρει να οσμιστεί αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε και σε επίπεδο δημοσιονομικό και να προχωρήσουμε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση σχετικά τώρα με το λεγόμενο κράτος δικαίου. Εμείς ήδη από τον Δεκέμβριο είχε γίνει δεκτή η έκθεση αυτή για το Rule of Law και από τότε δεν ακούσαμε τίποτα από το Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε στην διάθεσή μας για την διαπραγμάτευση θα μπορέσουμε με σοβαρό τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό. Thank you. Does the Commission want to intervene on... Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο για τα θέματα τα οποία τέθηκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσει να είμαι, να είμαι σύντομος από πλευρά τη ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσουμε την πολλή δουλειά και σοβαρή δουλειά την οποία έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το μελλοντικό ε, πολιετές και για τους ιδίους πόρους. Επίσης είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την άμεση ταχύτατη σύσταση της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου. Επί της ουσίας τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή της για το πολιετές δημοσιονομικό του 18 είναι μια σοβαρή βάση, σταθερή βάση για τη συμφωνία. Και αυτό de facto έχει αποδειχθεί άλλωστε από τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες είτε έχουν ήδη ξεκαθαριστεί είτε βρίσκονται σε επίπεδο τελικής διατύπωσης σχετικά με το πλαίσιο του 1,11% το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1,3% ενώ γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο πάρα πολλές χώρες μέλη θέλουν να μειώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιες ακραίες προτείνουν το 1 ακριβώς της 100. Σχετικά τώρα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ε, νέας Προέδρου, εδώ μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεων ανάμεσα στις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα εδώ. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής των προτάσεών σας θα πρέπει να ενταχθούν, να συμπεριληφθούν στις υπάρχουσες προτάσεις, οπότε θα χρειαστούν ε, λίγες τροποποιήσεις στόχων, επιμέρους και μόνο να αναφερθώ συγκεκριμένα σε τέσσερα θέματα τα οποία ήρθαν σε συζήτηση σήμερα, ευελιξία, ήδη πόροι, έκτακτες προβλέψεις και κλιματολογική αλλαγή. Σχετικά με την ευελιξία, υπάρχει ένα σαφής κίνδυνος το Συμβούλιο να προσπαθήσει να μειώσει το υπάρχον επίπεδο της ευελιξίας στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού. Είναι βασικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ευελιξίας που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι το παρόν σύστημα δημιουργήθηκε χάρη σαν ε, και στην αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του 2013. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργικό, δουλεύει καλά και έχει επιτρέψει στα ευρωπαϊκά όργανα να αντιμετωπίσουν σημαντικές κρίσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις ε, ε, από το 2014 και μετά. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας σχετικά τώρα τους νέους, με τους νέους ιδίους πόρους. Να μου επιτρέψετε να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Είναι πρώτη φορά για 22 χρόνια που έχω λάβει θετικά μηνύματα από το Συμβούλιο για νέους ιδίους πόρους. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό είναι θα έλεγα κάποια καλά νέα. Υπάρχει στήριξη λοιπόν και για τον ίδιο πόρο για τα πλαστικά και για το ETS υπάρχει μια κάποια στήριξη. Είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχουμε καταλήξει φυσικά ακόμα. Είμαστε μακράν μιας τελικής απόφασης. Απαιτείται, νομίζω, να εξετάσουμε και άλλες νέες δυνατότητες πέραν του αρχικού καλαθιού το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτά αναφέρθηκαν πολλά μέλη εδώ. Σχετικά τώρα με τις έκτακτες προβλέψεις. Ε, είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί ως ερώτημα προς τον Επίτροπο Χάν για την ακρόασή του. Ε, οπότε ο κύριος Χάν θα μας δώσει τις απαντήσεις. Να θυμίσω όμως ότι η ίδια η συνθήκη προβλέπει το πλαίσιο για τις έκτακτες αυτές ε, πιστώσεις, προβλέψεις μάλλον, ε, γιατί ε, η συνθήκη λέει ότι αν τυχόν δεν υπάρξει συμφωνία για το νέο δημοσιονομικό, όλες οι ισχύουσες ρυθμίσεις του προηγούμενου δημοσιονομικού συνεχίζουν να ισχύουν και για μετά το 2021. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο προβλέπει η συνθήκη. Πολλά μέλη επίσης αναφέρθηκαν στην ανάγκη να είμαστε πιο φιλόδοξοι στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι ο στόχος του 25% τον οποίο έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κλίμα είναι ένας στόχος φιλόδοξος, πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικός και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις προτινόμενες αλλαγές σε δημοσιονομικό επίπεδο και ιδιαίτερα την αυξανόμενη σημασία την οποία έχουν ορισμένες ε, τομείς κατά προτεραιότητα, πολύ σημαντικοί τομείς, αλλά που δεν έχουν ε, σε καμία περίπτωση σχέση με το κλίμα, όπως ασφάλεια, άμυνα, προστασία <clears throat> των συνόρων και Erasmus Plus. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις εδώ, σε κάποιες από τις προτάσεις ε, αφεαυτής μια αύξηση του Erasmus Plus θα μειώσει σαν παράδειγμα την, ε, τις προβλεπόμενες δαπάνες για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Το 25% εδώ νομίζω ότι είναι ένας στόχος επιτεύξιμος. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε με μία μικρή υπενθύμηση. Η σημασία του σεβασμού των αρμοδιοτήτων και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας είναι κάτι σημαντικό. Απαιτείται σύμφωνη γνώμη για το πολιετές, αλλά για τους ιδίους πόρους είναι συναπόφαση. Θα κλείσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει το διάλογο, αλλά σε αυτή τη φάση, στα πλαίσια της διαδικασίας, είναι στα χέρια της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εμείς σαν Επιτροπή θα συνεχίσουμε να παίζουμε το ρόλο διευκόλυνσης του διαλόγου και να συνεχίσουμε να απευθύνουμε εκκλήσεις για συνέχιση της σωστής συνεργασίας και για τακτικές επαφές και επικοινωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή ακούγοντας τους εισηγητές. Ας ακολουθήσουμε αντίστροφα τώρα την σειρά ο κύριος Φερνάντες για τους ιδίους πόρους. Αν κατάλαβα καλά, μόλον ότι δεν είναι πολύ καλά τα αγγλικά μου και σας ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη γι' αυτό, αν κατάλαβα καλά πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι θα κάνει περικοπές. Θα πρέπει τότε να γνωρίζουμε και ποιες περικοπές θα κάνει, έτσι δεν είναι, διότι αν μας λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έχουμε το τριπλάσιο ποσό για το Erasmus Plus, αλλά ότι θα πρέπει αυτό να προβλέπεται χωρίς να αυξηθεί το γενικό ποσό του προπολογισμού, τότε αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει ως εκθαύματος. Θα έχουμε μια θαυματουργή ευελιξία. Όχι, για μένα αυτό σημαίνει περικοπή. Περικοπή κάπου αλλού. Αν οι προτάσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν τηρηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Budget, δηλαδή ότι θα έχουμε το ίδιο επίπεδο προπολογισμού και μάλιστα ότι θα έχουμε και αυξήσεις, αυτό μας είπε, τότε ας μας πει ξεκάθαρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπονται τελικά περικοπές, πού θα γίνουν αυτές οι περικοπές. Εμείς ακολουθούμε τη μεθοδολογία της προσθετικότητος, δηλαδή και συμφωνεί με αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι λέει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να είναι σύμμαχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν λοιπόν τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας λέει ότι θα διατηρήσουμε τα ποσά, αλλά θα κάνουμε κάπου κάποιες αυξήσει, τότε είναι σαφές ότι θα κάνουν και κάπου περικοπές, έτσι δεν είναι. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται εύλογα αυτή τη στιγμή είναι πού θα γίνουν αυτές οι περικοπέ, μόνο ότι μπορώ να σας πω ήδη από τώρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να τις δεχθεί αυτές τις περικοπέ. Γιατί το ότι προσθέτουμε σημαίνει ότι προσθέτουμε καινούριου πόρου, όχι ότι κόβουμε κάπου αλλού. Λοιπόν, τίθεται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Μάρκε, τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό που είπε η συνάδελφος, η κυρία Γουαρδία Σαμπάλ, Σε ό,τι αφορά τις νέες προτεραιότητες, τα νέα προγράμματα, χρειάζονται πολύ απλά και καινούριο χρήμα. Και αυτό είναι για μένα το καθοριστικό στοιχείο. Όχι το πώς θα προσθέσουμε νέα στοιχεία, όπως είπε ο κύριο Φερνάντες, αλλά πώς θα μπορέσουμε να αναιρέσουμε τις προτάσεις σε ό,τι αφορά την περικοπή του προϋπολογισμού. Κύριε Τρέιλε, θέλετε να απαντήσετε μήπως σε αυτά που ακούσατε, σε αυτά που σας ρώτησαν ο κύριος Φερνάντες όλος ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές που μας κάνατε δεν έχω οποιαδήποτε εντολή για να επισέλθω σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας και να αναφέρω πιο πολλά στοιχεία. Σήμερα θα χρειαστούν κάποιες ε, τροποποιήσεις, αλλά εν ώψη και των ακροάσεων των μελλοντικών επιτρόπων δεν έχω να δηλώσω κάτι παραπάνω. Προφανώς όμως και σημειώνω το ερώτημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο ή μήπως ε, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η μηπως ολοκληρωσαμε τη σημερινη μας συνεδριαση σας ευχαριστω πολυ λεει η